Καλημέρα, συνάδελφοι. Σήμερα βρισκόμαστε σε τεράστια αίθουσα, γιατί πάντα είχαμε μεγάλη προσέλευση και δεν μας έφταναν και τα έντρανα, αλλά σήμερα φαίνεται ότι μας φτάνουν και μας περισσεύουν. Ναι, με καταλαβαίνετε, έχω ανάψει το μικρόφωνο. Και αυτό σίγουρα σχετίζεται με το γεγονός ότι δύο... έχει ανάψει το λαμπάκι στο μικρόφωνο, λέει η Πρόεδρος. Έχει ανάψει το φωτάκι στο μικρόφωνο, γι' αυτό νομίζω ότι λειτουργεί και η διερμηνία. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν είναι αθρώα η προσέλευση σήμερα, λέει η Πρόεδρο, σχετίζεται με το γεγονός ότι δύο ομάδε έχουν δύο έκτακτες ε, συνεδριάσεις. Η πράσινη στον ΙΜ και ε, το ΕΛΚ στη Μαδέρα. Τουλάχιστον κάποια από το ΕΛΚ, γιατί τα άτομα τα οποία μας ενδιαφέρουν από το ΕΛΚ είναι εδώ. Μας ζήτησε συγγνώμη και ο συντονιστής του ΕΛΚ, ο οποίος δυστυχώς ασθενεί. Να διατρέξουμε όμως την ημερήσια διάταξη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Έχετε λοιπόν τα έγγραφα στη διάθεσή σας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν προσθήκες για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Ωραία. Έγκρινεται λοιπόν όσο έχει η ημερήσια διάταξη. Να περάσουμε στο 2. Για την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 9 η Σεπτεμβρίου και της 23ης Σεπτεμβρίου. Όπως πάντα, αν μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης δεν έχω ακούσει οποιαδήποτε ένσταση σε ό,τι αφορά τα πρακτικά, θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί. Και άρα περνάμε στο 3 της ημερησίας διαταξής. Δεν έχω πολλά να σας ανακοινώσω. Αυτό που θα ήθελα να πω πριν από τις συζητήσεις είναι το εξής, ότι η συνεδρίαση η χθεσινή με την αντιπροσωπεία των Πολωνών συναδέλφων. Μεγάλη ομάδα ε, Πολωνών συναδέλφων που συμμετέχει στην Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονό και δεν το έχω δει σε, καμία, σε κανένα άλλο εθνικό κοινοβούλιο. Ασχολούνται πραγματικά εντατικά με τι επόμενε δημοσιονομικέ πρόπτικε και την ενδεχόμενη ε, αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση των πολιτικών. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε κανένα άλλο εθνικό κοινοβούλιο. Επί μια μισή ώρα λοιπόν συζητούσαμε και πολλοί Πολωνοί συνάδελφοι έλαβαν το λόγο, εξέφρασαν ασφαλώς και τις επιθυμίες τους. Θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη αυτή η εκδήλωση και συμμετείχαν ασφαλώς και κάποιοι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι τέτοιες συναντήσεις μπορούν να αποβούν πιο καρποφόρες από μεγάλες συναντήσεις όπου έχουμε προσκαλέσει όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Και έτσι έρχονται, ας πούμε, δύο εκπρόσωποι κάθε εθνικού κοινοβουλίου. Αυτό λοιπόν που έγινε χθες με έκανε να καταλάβω ότι εν μέρη Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την εργασία μας από το αν μιλάμε σε επίπεδο κυβερνητικό ή από όταν μιλάμε σε επίπεδο κοινοβουλίων. Ήταν πολύ χρήσιμη εμπειρία και θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετείχαν ε, συμμερίζονται την άποψη αυτή. Το επόμενο σημείο. Στους συντονιστές καταρτήσαμε το σχέδιο εργασιών μας, το οποίο λίγο πολύ έχει οριστικοποιηθεί. Φυσικά είμαστε ευέλικτοι, με τίθεται θέμα, αλλά έχετε λάβει πλέον τις ημερομηνίες, το σχέδιο των εργασιών μας, το πρόγραμμα των εργασιών μας, σε ό,τι αφορά το έτος 2011. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις. Αλλά φυσικά υπάρχουν και περιορισμοί. Πολύ απλά δεν γίνεται αλλιώς σε ορισμένες περιπτώσεις. Δύο φορές έχουμε ε, μια συνεδρίαση η οποία συμπίπτει με την Επιτροπή Αντιμετώπισης της Κρίσης και προχτές ε, προσωπικά ε, μίλησα με τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι τι να γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά και η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης ε, έπρεπε να λάβει υπόψη το πρόγραμμα εργασίας άλλων επιτροπών της Επιτροπής ε, Οικονομικών, για παράδειγμα, της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Εμείς φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη και της εργασίας της Επιτροπής Προϋπολογισμών και Ελέγχων του Προϋπολογισμού. Χρειαζόμαστε και διερμηνία και καταλαβαίνετε τέλο πάντων ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ιδιαίτερα επειδή θέλαμε να αποφύγουμε να διοργανώσουμε συναντήσεις σε πέμπτη απόγευμα, εφόσον είναι δυνατόν, και να αποφύγουμε και τις συνεδριάσεις στο Στρασβούργο. Δεν θέλουμε δηλαδή και συνεδριάσεις μια μισή ώρα πέμπτη απόγευμα. Θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας δυόμιση-τρεις ώρες στη διάθεσή μας. Γιατί ακόμα και σε δυόμιση ώρες, το είδαμε την προηγούμενη φορά, ε, δεν μας αρκούν σε πολλές περιπτώσεις, όταν θέλουν πολλοί συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Αν λοιπόν δεν έχετε αντιρρήσεις, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, θεωρώ λοιπόν ότι το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 ε, έχει εγκριθεί όσο έχει. Εν τω μεταξύ. Έστειλα και μία επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής όπου αναφέρω ότι καμία αντιπροσωπεία δεν έχει διοργανωθεί καμία αντιπροσωπεία και τέτοιες εκδηλώσεις από την Επιτροπή μας αλλά να το λάβουμε υπόψη ότι θέλουμε να έχουμε και μία έγκριση ad hoc σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι για να έχουμε μια τέτοια ευελιξία. Συμφωνήσαμε με τους συντονιστές. ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερο νόημα στο να διοργανώσουμε κάποια ταξίδι, κάποιες αντιπροσωπείες από την Επιτροπή μας. Ύστερα, επειδή το συζήτησα και με κάποιους συναδέλφους μετά την τελευταία συνεδρίαση, έγραψα μια επιστολή και προς όλους τους ε, επικεφαλείς όλων των επιτροπών και τους ε, διαβεβαίωσα ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με όλες τις επιτροπές και ότι θέλουμε να καταρτήσουμε, α, συγγνώμη, ότι θέλουμε να λάβουμε γνωμοδοτήσεις από τις επιτροπές τους, ωστόσο εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος, γιατί αν ε, λάβουμε μια ε, γνωμοδότηση τέλη Μαρτίου, πολύ απλά είναι πολύ αργά. Θα τις θέλαμε τις γνωμοδοτήσεις αυτές μέχρι τον Ιανουάριο, για να μπορέσουμε να τις εξετάσουμε. Διαφορετικά και τα μέλη τα οποία συμμετέχουν και σε άλλες επιτροπές θα μπορούσαν πάντα να μας μεταφέρουν το τι λέγεται και στις άλλες επιτροπές. Και να αντιπροσωπεύσουν και την ε, άποψη της ε, Επιτροπής. Άρα δια, διευκρίνησα ότι θεωρώ ότι οι πρόεδροι των Επιτροπών θα δώσουν την ευκαιρία στα μέλη τους να τους αναφέρουν την πρόοδο της Επιτροπής των εργασιών μας. Να μην αγνοούν τι γίνεται δηλαδή. Αυτές ήταν ε, οι ανακοινώσεις μου, οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Την προηγούμενη φορά και περνάμε τώρα στο 4 της ημερήσιας διάταξης. Ξεκινήσαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά να πραγματευόμαστε την έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου διευκρινίζεται, διευκρινίστηκε μάλλον την προηγούμενη φορά ποια είναι η θέση της Επιτροπής και μας βοήθησε αυτό ιδιαίτερα σε πολλά σημεία. Έχουμε και το σχέδιο εγγράφου του συναδέλφου Γκαρίγα. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη βάση επί της οποίας θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Και όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μας για το θέμα αυτό, ο συνάδελφος Σάλβαντρο Γκαρίγα θα καταρτήσει ένα σχετικά επίσημο έγγραφο εργασία το οποίο και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Δηλαδή, έχουμε καταρχάς το reflection paper στα αγγλικά, στην αγγλική γλώσσα και μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων λαμβάνοντας υπόψη και όσα έχουν υποθεί από τους συναδέλφους θα καταρτιστεί το σχέδιο το έγγραφο εργασίας και αυτό το έγγραφο εργασίας ε, θεωρώ εγώ προσωπικά αποτελεί την επίσημη άποψη της Επιτροπής μας, το οποίο θα διατεθεί και στο διαδίκτυο προκειμένου να μπορεί να το κατεβάσει όποιος ενδιαφέρεται. Την προηγούμενη φορά. Είχαν ζητήσει τόσο πολύ συνάδελφοι το λόγο που δεν μας έφτασε η ώρα και έχω ακόμα λοιπόν κατάλογο των ομιλητών που ήθελα να πάρουν το λόγο την προηγούμενη φορά για την έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Αλλά να πω αυτής εξ αρχή. και μάλιστα σας το ανακοίνωσα και εγγράφος ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο και τη μέθοδο εργασίας για την Επιτροπή μας. Δεν επιθυμώ πλέον να συμβεί αυτό που συνέβαινε και στο παρελθόν. Κάθε ομάδα, ανάλογα με το μέγεθός της, να ε, παίρνει το λόγο και να παίρνουν το λόγο οι συντονιστέ. Όχι, θέλω να υπάρχει μια πιο ευρεία συζήτηση και οι συντονιστέ. οι συντονιστέ σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα μέλη τη ομάδα του να κοιτούν, για παράδειγμα, ποιο έχει εξειδίκευση σε κάποιο θέμα. Και να μην χρειάζεται απαραίτητα να ζητούν το λόγο. να καταρτίζουμε έναν κατάλογο και μπορεί να υπάρχουν κάποια ειδικά θέματα και θα μου το λένε αυτό οι συντονιστέ από τον προτέρων ότι ο Χίψη είναι ο ειδικό εξ, εξ ονόματο από την ομάδα μα, ο οποίο μπορεί να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό, για να υπάρχει πιο μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων. Γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι αυτοί που θέλουν να πάρουν το λόγο, όχι μόνο τα πέντε τακτικά μέλη, αλλά και οι αναπληρωτέ ζητούν το λόγο. Και αν τελικά μαζεύονται 100 εισηγήσει, ε, πρέπει να βρούμε μία άλλη μέθοδο προσέγγισης. Και παράλληλα, το γεγονός ότι και εγώ μακρηγόρησα τώρα, να σας παρακαλέσω να είσαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. Γιατί πολλέ φορέ ε, τα καταφέρνουμε. Ξέρετε και στην Ολομέλεια τα καταφέρνουμε. Γιατί να μην είμαστε σύντομοι και εδώ. jetzt werden wir in die Ωραία λοιπόν, να συνεχίσουμε την συζήτηση της προηγούμενης ε, συνεδρίασης και να πω εξ αρχής ότι η πρώτη θα ήταν στον κατάλογο αγορητών η Ντανούτα Χίμπνερ. Αλλά, αλλά η Ντανούτα Χίμπνερ μας έχει αποστείλει γραπτά το, την εισήγησή της. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ λόγω της συνεδρίασης του ΕΛΚ στην Μαδέρα. Άρα λοιπόν δεν θέλει να πάρει το λόγο. Η Έστεν είναι η επόμενη στον κατάλογο αγορετών. Και το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται στο σημείο αυτό γιατί και αυτή είναι με το ΕΛΚ στη Μαδέρα. Και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σαμπάλ. Η Έντα Σαμπάλ. Γιούτα, σε ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι φαίνεται θα είμαστε σύντομοι γιατί είμαι πάρα πολύ αυτοί που ζήτησαν το λόγο αλλά δεν μπόρεσαν ε, δεν, θα μπορέσουν να τοποθετηθούν γιατί ανέλαβε και ο Σελβαδόρο το, το έγγραφο αυτό που θα αποτυπώνεται η θέση μας. Την τελευταία φορά πάντως που τα είπαμε, πάρα πολύ είχαν λάβει το λόγο όσον αφορά το, αυτή την, την έννοια της προσθέμενης αξίας και όντω ακούστηκαν ενδιαφέροντα αλλά και το έγγραφο περιέχει ενδιαφέροντα και αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί είναι το που εστιάζεται η ε, ο τόνος του έγγραφου δηλαδή, που δεν νομίζω ότι είναι ο πιο δόκιμος νομίζω ότι γι' αυτό το έγγραφο προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε αποπειρώμεθα να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη της ε, Ευρώπης κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να διαπνέει αυτή την προβληματική γιατί έχει δείξει και με το παραπάνω η Ευρώπη ότι δικαιολογείται η ύπαρξή της άρα δεν χωρεί συζήτηση για αυτό το θέμα. Πάντως αυτό που μου φαίνεται εμένα λογικό είναι το να δούμε τι θα γίνει με την προστέμενη αξία των πολιτικών. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Όταν κάτι τέτοιο χαράζεται, αποφασίζεται και σε την Ευρώπη και παντού, εθνικά, περιφερειακά κλπ. Ε, τότε ε, είναι πάρα πολύ ε, σωστό το να συζητείτε η αξία, κάτι το οποίο ανέκαθεν γινόταν και γι' αυτό νομίζω ότι η αναγκαιότητα του να συζητήσουμε την προστεμένη αξία είναι το ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες πολιτικές θέλουμε να χαράξουμε, ποιες θέλουμε να υλοποιήσουμε και από αυτές ε, ποιες θέλουμε να ε, προχωρήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιε να έχουν χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και τα λέει στο έγγραφό του ο Σαλβαδόρο. Το θέμα δεν είναι να κάτσουμε να αποτιμήσουμε τη διαχείριση, ε, της εξοικονομήσεις δαπανών, την αποτελεσματικότητα. Αυτό που θέλω να δούμε είναι η προσθεμένη αξία. Δεν είναι κάτι μόνο ποσοτικά αποτιμητέο. Πολλές φορές είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Ε, και το λέγεται το έγγραφο ότι ο πλευρά ε, ποσοτική δεν γίνεται, δεν πρέπει να καθόμαστε να, να, να, να ακριβώς τι έγινε. Αυτό που χρειάζεται είναι η ε, προσθέμενη αξία, η, η ειρήνη. Αυτό είναι το πιο αποφασιστικό. Επομένως, όσον αφορά τα διάφορα επίπεδα ε, αποφάσεων, να δούμε ποιο είναι το πιο προτιμητέο και αυτό θα πρέπει να δούμε, ότι οι πολιτικές που θα πρέπει να ασκηθούν θα πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο θα αποφασίζονται και αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε από πλευρά ευρωπαϊκής και από πλευρά προϋπολογισμού της Ένωσης, από πλευρά της προστιθέμενης αξίας, από πλευρά αυτών των πολιτικών και σας ε, προαναφέραμε ότι αυτό ήδη έχει γίνει και γι' αυτό νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ξαναμελετήσουμε αλλά όχι έχοντας αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιολόγησης αλλά για να επιφέρουμε βελτιώσεις και για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα και να σκεφτούμε τι μπορούμε να επιφέρουμε σαν βελτιώσεις, ας πούμε στην πολιτική της συνογής. Ε, προφανώς οι χώρες οι οποίες ε, ε, είναι επιλέξιμες βεβαίως και για αυτές είναι κάτι το καλό και υπάρχει προσθεμένη αξία, αλλά και οι χώρες ε, δωρητές και αυτές έχουν προσθεμένη αξία. Επομένως, η ανάλυση δεν είναι σε σχέση με το ποιος πήρε και ποιος έδωσε, αλλά ξεκίνησε αυτή η ιδέα σαν μια συμφωνία μεταξύ των περισσότερων και των λιγότερων αναπτυγμένων, τόσο ώστε να φτάσουμε σε ενιαία αγορά. Η ΚΑΠ είναι επίσης ένα κλασικό παράδειγμα προστιθέμενης αξίας. Είναι αυτονόητο ότι πρόκειται να έχουμε κοινωτική πολιτική, ε, και, ατομικά και συλλογικά, αλλά όλες οι χώρες θέλουν μια τέτοια αγροτική, γεωργική πολιτική, κοινή για τους 27. Μία κοινή πολιτική. Είναι αυτό πιο λογικό, είναι πιο επικερδές παρά το να έχουμε 27 διαφορετικές γεωργικές πολιτικές. Τι σημερινή μέρα δεν νομίζω ότι κάθεται κανένας να λέει ότι δεν χρειάζεται ε, κοινή δαπάνη, κοινή, κοινό συντονισμό, αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, αυτά πάντοτε λέγαμε ότι θα χρειάζεται να, να βελτιώσουμε τα πράγματα, ε, χρειάζεται να την αναβαθμίσουμε σε κάθε επίπεδο. Πρόκειται για μια πολιτική που θα πρέπει να συνεχιστεί, να την επεξεργαστούμε περισσότερο και αυτό που σήμερα συζητείτε, δηλαδή η εξωτερική δράση, η εξωτερική πολιτική. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα και των Ευρωπαίων αλλά και των χωρών της Ευρώπης ότι θέλαμε να υπάρχει μια τέτοια κοινή εξωτερική πολιτική. Όμως για το μέλλον υπάρχουν αυτά τα πράγματα που τώρα πέφτουν σαν ιδέες, θα τα επεξεργαστούμε, θα προχωρήσουν στο μέλλον και άρα να αναζητήσουμε και άλλες νέες πολιτικές. Διότι χρειάζεται ένα σλόγγαν, ένα light ένα σύνθημα. Εποδός, να, να είναι μια βιώσιμη ε, μια Ευρώπη βιώσιμη από πλευράς οικονομικής, κοινωνικής, αλλά και βιώσιμη από πλευράς περιβαλλοντικής. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κάτσουμε και να αξιολογήσουμε ποιε είναι οι πολιτικέ που θα πρέπει να ασκήσουμε και ποιε πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και να συντονίσουμε από πλευρά τη Ευρώπη. Έχουμε και όλα αυτά τα, τα μέσα οικονομική διακυβέρνηση υποδομές, ενέργεια, μεταφορές, καινοτομία. Όλα αυτά καλύπτονται από την υπόθεση στρατηγική 2020 που και θα συζητήσουμε. Από πλευράς κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύη, ε, καταπολέμηση περιθωριοποίησης, προστασία του, κλίματος, της αλλαγής του κλίματος και καταπολέμηση εξωτερική δράση, όλα αυτά τα συζητήσουμε, αλλά πάντοτε, όπως σας έλεγα, ο στόχος είναι να εξεταστεί ε, το τι έγινε, αλλά και στο μέλλον τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Και ε, είναι κάτι αυτό που εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευλάς πολιτικής, αλλά και από πλευράς δημοσιονομικής. Και αυτό είναι και η δουλειά μας στην Επιτροπή να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Πάουλσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ολλανδικά. Ολλανδικά. Νομίζω, αν με επιτρέπετε, να σας αναμίξω δύο έγγραφα προβληματισμού που έχετε υποβάλει. Αφενός για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, νομίζω ότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, να ποσοτικοποιήσουμε την αξία αυτή, δηλαδή τι αξίζει οικονομικά να υλοποιηθεί είτε πολιτικά, αν όμως το δούμε είτε πολιτικά είτε κοινωνικά είναι πολύ δύσκολο. Για παράδειγμα η αγροτική πολιτική όπου βέβαια χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε τα τρόφιμα που παράγει η αγροτική οικονομία είναι όμως δύσκολο να ζυγιστούν τα διάφορα στοιχεία που συναπαρτίζουν την αγροτική πολιτική. Ο καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας, το καθαρό νερό, αυτά δεν είναι ωστόσο μετρήσιμα. Στον προϋπολογισμό τώρα νομίζω ότι είναι λάθος η αφετηρία του εδώ στην Ευρώπη. Μα προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε οράματα τα οποία ίσως είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στην επόμενη ζωή. Οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένη. Ας είμαστε λοιπόν όριμοι να αντιληφθούμε ποια πράγματα αποτελούν μοναχά οράματα και ποια πράγματα είναι η πραγματικότητα. Ότι έχουμε περιορισμένους πόρους. Να κατανοήσουμε ότι στο μέλλον δεν μπορούμε να έλκουμε τον προπολογισμό αυτό προς πάσα κατεύθυνση ώστε να προσαρμοστεί στα οράματά μας. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε σωστή κατανομή των κονδυλίων που διαθέτουμε, να καταφέρουμε να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Έχουμε λιγότερους πόρους και περισσότερες ανάγκες. Άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους και να χρησιμοποιήσουμε κάθε τι που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να δημιουργήσουμε μια προσθέμενη αξία. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Να θέσουμε στόχους και στόχους οι οποίοι μάλιστα να είναι μετρήσιμοι, δηλαδή να μπορούμε να μετρούμε την πρόοδο που κάνουμε προς την επίτευξή τους. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Καλφίν, τελευταίος από τον κατάλογο που είχε μείνει από την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σημαντικό είναι να λεχθεί και νομίζω να συνεχίσουμε και στο μέλλον την συζήτηση αυτή ότι δεν πρέπει να λησμονούμε δύο ιδιαιτερότητες του κοινοτικού προϋπολογισμού. Πρώτον είναι δημόσιος προϋπολογισμός με δημοσίους πόρους. με διαφορετικές βάσεις από ό,τι για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Όταν μιλούμε για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα μέσα, με λιγότερους πόρους, Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και βέβαια και τι θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό από τον φορολογούμενο. Όταν λοιπόν μιλούμε για θέματα που έχουν σχέση με προστιθέμενη αξία, αυτά που αρχίσαμε να συζητούμε την προηγουμένη φορά δηλαδή για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ας μιλήσουμε τα εξή. Πρώτο, δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι ο κοινοτικός προπολογισμός στα πλαίσια τα σημερινά, ένα περίπου της 100 του ΑΕΠ των χωρών μελών, θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα με τον τρόπο που αναμένει ο κόσμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε λοιπόν θα πρέπει θα πρέπει να καταστρώσουμε μια φιλόδοξη, φιλόδοξη πολιτική ατζέντα και μετά να ψάξουμε να βρούμε τους πόρους, είτε θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ατζέντα στους πόρους. Η ιδέα του να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα μου αρέσει και εμένα, αλλά κάθε βέβαια ε, προπολογισμό θα πρέπει να διαθέτει αποθεματικά για να μπορεί να κάνει κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να ε, ασκήσουμε νέες πολιτικές, να μπούμε σε νέους τομείς πολιτικής, μοναχά με τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε από αποτελεσματικότερη χρήση των υφισταμένων πόρων. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν και ποιοι είναι οι πόροι του προϋπολογισμού. Δεύτερο, το, ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός έχει και μια διαφορά από τις εθνικές. Ότι δηλαδή μπορεί να παίξει στην συμπληρωματικότητα με τις εθνικές πολιτικές. Μπορούμε να αναζητήσουμε λοιπόν την προστιθέμενη αξία με τη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού όταν τον συνδυάσουμε σωστά με συντονισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές και τις δαπάνες στο εθνικό επίπεδο. Και εδώ έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη το γεγονός ότι το έργο μας σχετίζεται με αυτό των εθνικών βουλών. Και βέβαια μέσα στο πλαίσιο των όσων κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια για την εποχή μετά την κρίση, μετά το 2013. Και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει καλύτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ό,τι δεν μπορεί να γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να γίνει στο εθνικό. Εδώ λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένα πού μπορεί να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. χωρίς να επεκτείνουμε τη συζήτηση σε άλλα θέματα ενδιαφέροντα μένα, αλλά όπου δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Ακόμα δεν έχουμε τις απαντήσεις από την συζήτηση αυτή. Μέχρι τώρα έχουν τεθεί ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, ακούσαμε ενδιαφέρουσες γνώμες, αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε να συνεχιστεί το έργο της Επιτροπής μας, θα πρέπει να βρούμε και απαντήσεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικότερα για την εξυπηρέτηση των στόχων και πώς μπορούμε να συντεριαστούμε με τις εθνικές ε, πολιτικές και ποιες είναι εκείνες που δεν μπορούν να γίνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το άλλο είναι το δεύτερο έγγραφο για το 2020 την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 το οποίο υποβάλλεται σήμερα οι ερωτήσεις είναι, υποθέτει δηλαδή το έγγραφο, είναι σημαντικές. Πρέπει να τις συζητήσουμε. Ορισμένε ορισμένες εξ αυτών δέχονται προφανείς απαντήσεις. Άλλες θα λάβουν διαφορετικές απαντήσεις από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Αλλά αυτό που θα πρέπει να είναι η καθοδηγητική ιδέα όταν μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 και του τι μπορεί να πράξει ο προπολογισμό τη είναι το εξή. Πρώτο, δεν μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε ολόκληρο τον προπολογισμό. Δεν θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή μετά το 2013. Όλες οι πολιτικές οι οποίες υφίστανται μέχρι τώρα μπορούν να βελτιωθούν, μπορούν ίσως και να αναθεωρηθούν, αλλά είπα να επανεξεταστούν. αλλά δεν μπορεί να είναι ένα το προπολογισμό του 2013, διότι όπω λέει και το έγγραφο, δεν καλύπτει τα πάντα στην, Ευρωπαϊκή, στην, Ένωση, στην ε, ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπαίνουν στο 2020 και δεν χρειάζεται. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποιοι είναι οι πόροι που μπορούμε να διαθέσουμε στις ε, προτεραιότητες, ε, να διαθέσουμε πόρους σε αυτές και τι μπορούμε να ταπανίσουμε για να τα επιτύχουμε αυτά. Πάλι εδώ τίθεται το θέμα του συντονισμού με τις εθνικές πολιτικές και είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε μονάχα στις 7 προτεραιότητες γιατί εκτός από τις σημαντικές τις flagship initiatives υπάρχουν και άλλες για την Ευρώπη του 2020. Πάλι θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο αφού μιλούμε για θέματα ευρωπαϊκού προορισμού. πώς καλύπτονται αυτές τις προτεραιότητες. Επίσης, να είμαστε πιο φιλόδοξοι για την εξισορρόπηση μεταξύ των προτεραιοτήτων του 2020, πρόσθετων προτεραιοτήτων και της διατήρησης κάποιου περιθωρίου για την επόμενη περίοδο. Γιατί αν εξετάσουμε το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα, κινδυνεύουμε να εξαντλήσουμε όλα τα αποθεματικά, όλα τα περιθώρια, λόγω των όσων εμφανίζονται μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν μεγαλύτερη ευκαμψία θα πρέπει να συνδυαστεί και μια προσπάθεια να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε τις προτεραιότητες. Μιλώ με γενικό τρόπο γιατί είναι και γενικές οι ε, ιδέες που περιλαμβάνει το έγγραφο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για το πώς μπορεί να βρει απήχηση η Ευρώπη του 2020 στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η πρόεδρος Ζήτα Χάουκ. Ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο μέρος της παρέμβασης του Κύριο Κάλφιν θα τον βάλουμε εκεί στην αποδοτικότητα. Γιατί μίλησε ταυτόχρονα και για ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και για Ευρώπη 2020. Στην αρχή όμως άκουσα κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζω να το άκουσαν καλά και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Υπουργών. Διότι η αξίωση όταν επινοούμε νέες πολιτικές ή νέα καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει και η απαραίτητη χρηματοδότηση. Αυτή η αξίωση είναι παλαιά, αλλά το Συμβούλιο πρέπει να την ακούσει, διότι το Συμβούλιο είναι αυτό που έρχεται κάθε τόσο με καινούργιες πολιτικές. Τώρα, για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Υπάρχουν ακόμα τρει που ζήτησαν το λόγο. Αντρεάσεν, Πόρτα. Α, μια στιγμή. Πρώτα ο Αλέξανδρος Άλβαρο μετά Αντρεάσεν, μετά Μιγκελ Πόρτας και θα ακούσουμε μετά τη σύνοψη του εισηγητού. Αλεξάνδερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω γιατί είπαν πολλά ήδη συναδελφοί μου. ο κοινοτικός προϋπολογισμός ακόμα και αν έτσι το βλέπουν ορισμένες ε, χώρες μέλη δεν είναι καθαρά συγχρηματοδοτικός μηχανισμός για εθνικά έργα γι' αυτό και δεν συμφωνώ απόλυτα με τον Καλφίν σε ό,τι αφορά τους εθνικούς προϋπολογισμούς εκεί όπου μπορεί να γίνει και πέραν των ορίων ορισμένων έργων, αυτή η συνεργασία είναι σωστό να γίνεται αυτή η συσχέτιση. Όταν όμως μιλούμε για μια εξίσωση προτεραιοτήτων του κοινοτικού προπολογισμού με εκείνους των εθνικών, τότε η συζήτηση είναι διαφορετική. Μιλούμε για ένα είδος streamlining της ε, ευρωπαϊκής κοινοτικής πολιτικής με τις εθνικές. Δεν νομίζω ότι όμω καμία από τι 27 χώρε μέλη σκέφτεται κάτι τέτοιο για την ώρα. Εάν το θέλουμε εμεί πρέπει να σκεφτούμε πώ θα δημιουργήσουμε του ε, μηχανισμού αυτού και πώ θα συνδυάσουμε τι προσπάθειε μα με εκείνες της ε, Κομισιόν. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται πρώτα-πρώτα ο συσχετισμό αυτό και με ποιο τρόπο τον καθορίζει ο προπολογισμό. Τώρα, το σημαντικό είναι και η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, ίσω σα φανεί γενική η παρατήρηση αυτή, Εκεί δηλαδή όπου μπορούμε εμεί να λειτουργήσουμε καλύτερα και από ότι μια εθνική χώρα, μια, συγγνώμη, μια χώρα μέλος μόνη της. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Όπου δηλαδή το σύνολο αποδίδει καλύτερα από τα μέρη. Εκεί λοιπόν λειτουργεί καλύτερα η Ευρώπη. Όταν έχουμε best practices, για παράδειγμα στην έρευνα και ανάπτυξη να δούμε πού μπορούμε ε, να δημιουργήσουμε κέντρα υπεροχής, να προσφέρουμε κατάλληλες συνθήκες εργασίας, εργασίας στους ερευνητές μας και ούτω καθεξής. Και αυτά πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ευτυχώς που στην παρούσα Επιτροπή μπορούμε να συζητήσουμε τέτοια πράγματα. Πού ακριβώς έγκυται οι προτεραιότητές μας ασφαλώς δεν είναι το Άγιο Δισκοπότηρο η ε, Ευρώπη του 2020. Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να λοιπόν να βρεθεί ένας... Έχουμε όμως το πρόβλημα πάντοτε, το είδαμε αυτό και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, ότι δημιουργούμε νέες προτεραιότητες, νέους στόχους, αλλά μετά όχι, μην θίξετε τον αγροτικό προϋπολογισμό, λένε οι μεν. οι άλλοι μας λένε μην θίξετε τα διαφθορτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Άλλοι, όπως εγώ, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα όσα έχουμε και ταυτόχρονα κάνουμε καινούργια πράγματα, τότε θα μας ρωτήσει το Συμβουλίο και δικαίω, μα πώς το βλέπετε το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι ο κοινοτικό προπολογισμό πρέπει να συνεχίσει να είναι ισοσκελισμένος και να δούμε πώ θα οργανώσουμε τι προτεραιότητε ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη με εύκαμπτο τρόπο και οι έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι που δεν συμμετέχουν στη δική μας Επιτροπή ή την Επιτροπή Κρίσεως ή Προϋπολογισμών κάπου σκέφτονται ότι ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναλάβει και χρέος. Θα μπορούσε να δανειστεί δηλαδή. Ευρωομόλογα δηλαδή εν προκειμένου. Εγώ νομίζω ότι είναι πραγματική ευλογία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δικαιούται να κάνει χρέη. Τα βλέπουμε, βλέπουμε την κατάσταση των εθνικών προϋπολογισμών. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν στις αρχές δεκαετίας του 80 είχαν πει τότε οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων μπορούμε να κάνουμε και χρέη. Θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση σήμερα. Θα είχαμε φτάσει τώρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητούμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας καλύψει. Κάπου πάει να σηκώσει το κεφάλι του το φάντασμα αυτό και εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες και να έχουμε ε, το ευρωπαϊκό αυτό πνεύμα στον προπολογισμό πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε και κάποια ταμπού. Δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, λέει η Ιούτα Χάουκ, ότι όλοι οι πολιτικοί δηλαδή απαιτούν προστασία των κεκτημένων, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν είναι η ιδέα συνολικά του Κοινοβουλίου. Έχω μιλήσει με διάφορες χώρες μέλη και τα ίδια είδα, είδα από όλες τις χώρες μέλη. Η καθεμία κάτι διαφορετικό βέβαια, γιατί για κάθε μία είναι διαφορετικά πράγματα σημαντικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ακριβώς λοιπόν το ίδιο συμβαίνει εκεί. Η κυρία Αντρεάσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω το εξής, ότι το έγγραφο του Σαλμαδόρα αποτελεί ένα έγγραφο περισυλλογής, αν θέλετε, ένα reflection paper και τίποτα παραπάνω ούτε θα μπορέσει να καταστεί κάτι παραπάνω, γιατί πολύ απλά λείπει κάτι πολύ βασικό στην ανάλυση αυτή. Η ενδιάμεση αναθεώρηση. Όσο, όσο την έχουμε στην διάθεσή μας, δεν θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και ε, πραγματικά δεν είμαι βέβαιη ποια είναι, ποιο είναι το καθήκον της Επιτροπής αυτής. Το είπα αυτό γιατί συζητάμε και τον ε, προϋπολογισμό για το 2011 επί του παρόντος. Μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό φόρο, νέους, ε, νέους ίδιους πόρους και ποια θα είναι η κατάσταση με, τα, με τις δαπάνες στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μία ε, αντίθεση μεταξύ του έργου των δύο επιτροπών και θα ήθελα να διευκρινίσουμε το καθήκον της Επιτροπής μας. Ύστερα, να πω το εξή. Για να καθορίσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα τελευταία χρόνια πόσο, κατά πόσο ήταν αποδοτικό ο ευρωπαϊκό κοινωνικό προπολογισμό. Γιατί δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό ο τρόπο με τον οποίο ε, προγραμματίζουμε και καταπτύζουμε τον προπολογισμό. Γίνονται πολλέ μεταφορέ για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που ξεμένουν σε πολλές γραμμές του προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε αυτό για να καθορίσουμε το πού μπορεί να βρεθούν οι πόροι χωρίς να σκεφτόμαστε περί ευρωπαϊκών φόρων. Και το τελευταίο που ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. Είναι δύσκολο να σκεφτόμαστε το ποια θα είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στα κράτη-μέλη. Γιατί στην τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη μπορούν να το κρίνουν μόνο αυτό. Αν δεν συνομιλούμε λοιπόν με τα εθνικά κοινοβούλια, με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, συμφωνώ με τον κύριο Κάλφιν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, δίωδος επικοινωνίας με τα εθνικά κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Μιγγέλ. Eh, Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω να σας πω να σας εξηγήσω κάποια σκέψη μου σε σχέση με αυτά τα οποία ακούσαμε γιατί ακούσαμε ε, το, τα σχέδια με τον προπολογισμό, το τι θα γίνει στο μέλλον, όταν ενδεχομένως έχουμε πιο περιορισμένους πόρου διαθεσή μα για να δούμε. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα και διευρύνονται δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας και για αυτό το λόγο ε, ε είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και στις ε, χώρες μας σε σχέση με τις αρμοδιότητες των ε, περιφερειακών ή εθνικών ή, περιφερειακών, ή τοπικών περιφερειακών αρχών σε σχέση με τα κονδύλια το οποία έχουν Πάντως, κάθε υπηρεσία, κάθε θεσμικό όργανο, αν δεν έχει πώς διάθεσή του, προσπαθεί να νομοθετήσει όλο και περισσότερο. Και αντιστρόφως. Επομένως προσπαθούν νομοθετικά να λύσουν τα προβλήματα όταν δεν μπορούν να τα λύσουν με χρήματα που στη διάθεσή τους. Είναι αυτό ένα έθιμο, μια παράδοση πάρα πολύ κακή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ισχύει. Έχουμε τώρα μια παραπάνω δυσκολία. Χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ο μελέτα χωρίς αυγά δεν γίνεται επομένω. Θα καταλήξουμε να έχουμε λιγότερη Ευρώπη. Και λιγότερη ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Γι' αυτό σας ρωτώ, συνάδελφε, για να δούμε. Σε ποιους τομείς πολιτικής θέλουμε λιγότερη Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει βιομηχανική πολιτική, αλλά έχει 14 προγράμματα που αφορούν τη βιομηχανία. Ο, το, ιδεα σχέση κόστους οφέλους αυτών των 14 προγραμμάτων θα πρέπει να αναλυθεί. Είναι αρνητική η σχέση. Και τι θα κάνουμε, θα τα κόψουμε αυτά τα προγράμματα ή θα προσπαθήσουμε να αποκτήσει βιομηχανική πολιτική, αρμοδιότητες βιομηχανικής πολιτικής Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, τι πρέπει να συζητηθεί. Άλλο παράδειγμα, η στρατηγική για την ενιαία εσωτερική αγορά θα πρέπει να έχει ως στόχο την ομογενοποίηση, την εναρμόνιση όσον αφορούν, όσον αφορούν τα είδη διατροφής. Να ποιο είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με ε, κάποια πιάτα τοπικά, περιφερειακά. Ναι, να έχουμε λιγότερη Ευρώπη, τόσο ώστε να προστατεύσουμε τη διαφορά. Αυτά τα διαφορετικά προϊόντα, τα οποία έτσι διαφορετικά αν έχουν πρόσβαση στην αγορά. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας δείξω ότι η προβληματική δεν είναι καθόλου απλή. Πάντως, πέραν αυτών, στην επόμενη οκταετία, δεκαετία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η απόκληση που τα σημειώνεται μεταξύ των χωρών που έχουν πλεόνασμα και των χωρών που έχουν έλλειμμα. Και μιλώ για το εμπορικό ισοζύγιο. Να, ποιο είναι το πρόβλημα. Τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Η Καλιφόρνια βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, ξέρετε. Όμως ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός αντιστοιχεί στο 20 και του ΑΕΠ. Εμείς θα κάνουμε το 2020. Εμείς θα έχουμε προϋπολογισμό που θα είναι λιγότερο το 2% του ΑΕΠ στην Ένωση. Τι θα κάνουμε. Μήπως θα πρέπει να προχωρήσουμε προς λιγότερη Ευρώπη. Αυτό θα κάνουμε. Γιατί να. Να θα γίνει το 2010. Ε, Ευχαριστώ, Κίνγκα Γκέντ, Και μετά να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για να, να κάνει μια σύνοψη. Ευχαριστώ. Αν έχουμε λίγο χρόνο στην διάθεσή μας, νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την γραμμή αυτή. Συμφωνώ με όσους είπαν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλα θέματα πρωτού κοιτάξουμε ε, θέματα ειδική πολιτικής. Να κοιτάξουμε καταρχάς πώς οι ευρωπαϊκή πόροι για την αντιμετώπιση της κρίσης ε, είχαν αποτέλεσμα, βοήθησαν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την ε, κρίση και με βάση αυτό μπορούμε να κοιτάξουμε αν θέλουμε πιο πολύ ή πιο λίγη Ευρώπη για το μέλλον. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κρίση θα τελειώσει σε κάποια χρόνια και θα υπάρχει ανάκαμψη της οικονομίας σύντομα και τότε θα τεθεί το ερώτημα το κατά πόσο θα θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη και το πώς θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο πλαίσιο. Είδαμε ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης έχει περιοριστεί σημαντικά. καιρός λοιπόν θα ήταν να πάρει μια νέα όθηση του κατά πόσο θέλουμε πιο πολύ ή πιο λίγη Ευρώπη. Αυτό φυσικά αποτελεί ένα θέμα το οποίο υπησέρχεται σε κάθε συζήτηση. Αν θέλουμε πιο πολύ Ευρώπη και όλο και πιο πολλούς πόρους για την Ευρώπη, Αυτό φυσικά αποτυπώνεται και στις συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής και αναζητώντας ε, νέους πόρους, τίθεται φυσικά και πάντα το θέμα της αποδοτικότητας. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί εκ νέου με έναν πιο ομόφωνο τρόπο. Και ανακύπτει λοιπόν και το επόμενο ερώτημα, πώς θα μπορούσαμε δεχομένως να διαθέσουμε αυτούς τους επιπλέον πόρους και πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, να συλλέξουμε και άλλους πόρους. Κάθε φορά λοιπόν που τίθεται το θέμα του κατά πόσον θέλουμε πιο πολύ ή πιο λίγη Ευρώπη, τελικά η συζήτηση καταλήγει στα θέματα αποδοτικότητας. Και διαπιστώνω ότι σε κάποιους πολιτικούς τομείς θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν περαιτέρω περικοπές, γιατί δεν θα απέβαινε αυτό προς όφελος της αποδοτικότητας. Εκ παραλλήλου είναι σημαντικό να είμαστε σε διαρκή επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια και να υπάρχει μια προσαρμογή της πολιτικής, γιατί υπάρχει έλλειψη αποδοτικότητας λόγω έλλειψη εναρμόνιση. και αυτό προέκυψε με σαφήνεια χτε ε, κατά τη συζήτηση με τους εκπροσώπους του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Σαλβαδόρ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του αδέλφου όλου που έλαβαν το λόγο με όσα είπαν έδειξαν ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς ε, κατόπιν ε, το τόσο συζητήσαμε τελευταία φορά στο Στρασβούργο. Ε, τώρα πάντως πάρα πολλοί κόσμος έλειψε λόγω της γενικής υπηρεσία στην Γαλλία αλλά και το ίδιο ισχύει και σήμερα που, που λείπουν τόσοι συνάδελφοι εκτός Βρυξελών και ας Ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα συνεδριάσει η ΣΟΥΡΕ, η Επιτροπή μας, θα έχουμε ευρύτερη συμμετοχή. Πάντως, βούκαν τον πολλό του ΕΦ και ευχαριστώ για την ποιότητα των ε, εισηγήσεων του συναδέλφους και όλα αυτά τα οποία είπανε πρόκειται να τα εντάξω στο κείμενο το οποίο θα προκύψει κάποια στιγμή. ήδη. Ξέρετε ότι αυτέ οι πρώτε μας συνεδρίε αφορούν αυτό το έγγραφο μελέτης, το οποίο θα είναι βάση για συζήτηση. Και κάποιε μυθέ δεθούν και όλε αυτέ οι νέε ιδέε, ε, ε, όλων όσων έχουν κάποιε ιδέε, όλων όσων έχουν κάποιες γνώσει γνώσεις, όσον αφορά τις δημοσιογενεί προοπτικέ, αλλά και τον ε, ε, προπολογισμό. Όσον αφορά από αυτά που άκουσα σήμερα συγκεκριμένα, έχω να σα πω ότι ε, βασικά θέματα είναι το, αυτά τα οποία είπαμε στο Στρασβούργο. Δηλαδή, πόση Ευρώπη θέλουμε. Έχουμε την διαδρομή των τελευταίων ε, ετών με τις δημοσιονομικές προοπτικές και τους προϋπολογισμούς τους αντίστοιχους που μας δείχνουν ότι θέλουμε να εμβαθύνουμε για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και αντιστοίχως ο κοινοτικός προϋπολογισμός να γίνει πιο φιλόδοξος. Γι' αυτό και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούμε σε κάποιες ιδέες, σε κάποιες πολιτικές που δεν έχουν πάντα την αναγκαία πρικοδότηση. Πολλές φορές έχουμε κάποια προγράμματα φιλόδοξα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ σημαντική προστιμένη αξία. Όμως δεν υπάρχει αναγκαία χρηματοδότηση. μεταφορές πόρων από το ένα κονδύλιο στο άλλο, τη μία γραμμή προτιμού στην άλλη. Και πάρα πολλές φορές επομένως οι στόχοι δεν υλοποιούνται για αυτούς τους λόγους. Γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο πρώτο γύρο συζήτησης και να δούμε πόση Ευρώπη θέλουμε και κατά πόσο γίνεται να υπάρξει χρηματοδότηση με νέους πόρους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να εμβαθύνει για αυτό τον προβληματισμό πόσα προγράμματα σήμερα τρέχουν χωρίς να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση. Αν κάπου λείπει η κρίσιμη μάζα σε κάποιο πρόγραμμα. Όπως και είπε και ε, σαν Δεν υπάρχει κρίση μάζα, τόσο ώστε να υπάρξει κάποια συνέπεια πραγματική. Μήπως ε, πιο σωστό είναι να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα, πιο λίγα προγράμματα. Και το ίδιο ενισχύσει και με τους στόχους και με τους πόρους. Τα είπαμε και στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Έχουμε και εκεί μια εισήγηση να κάνουμε όσον ε, αφορά τους ιδίους πόρους. Και εδώ έχουμε τον κύριο Ντεχάνε. Ε, τον έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ντεχάνε στην Επιτροπή Σούρη για το τι θα γίνει με τους ιδίους πόρους, κατά πόσον μπορούν να αυτοί να μας ε, συμβάλλουν τόσο ώστε να προχωρήσουμε σε κάποιες άλλες μελλοντικές δημοσιομικές προοπτικές. ποια διάσταση θα έχουν τα πράγματα, τι θα γίνει με τον προπολογισμό. Όπω είπε και ο Σύνδεφο Πόρτα, πάμε για το 1 2% του προπολογισμού σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ. Εγώ θα βασιστώ πάντω ε, στην ε, απόφαση για του ιδίου πόρου. Εκεί όπου ορίζονται τα όρια, ορίζεται το τι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον προπολογισμό. Αυτή είναι η πραγματική βάση στη σημερινή συγκυρία μέχρι να υπάρξει κάποια απόφαση που θα αλλάζει τις δημοσιονομικές προοπτικές. Αν με ρωτήσετε για τις διαστάσεις του προπολογισμού του κοινοτικού θα σας πω ότι ναι, σήμερα δεν είναι αρκετός, θα ήθελα να είναι αυξημένος ο προπολογισμός αλλά πρέπει να είναι ρεαλιστής. Σήμερα έτσι έχουν τα πράγματα και άρα στο μέλλον θα δούμε κατά πόσο θα αλλάξει η σχετική απόφαση ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να ρίξουν περισσότερα χρήματα στον κοινωτικό προπολογισμό. Πάντως, η σημερινή τάση όπως ξέρετε είναι αντίθετη γιατί πάρα πολλές χώρες στο Συμβούλιο προκοιτάνε πώς θα ρίξουν όσο γίνεται λιγότερα χρήματα στον προπολογισμό. Να επομένως τι γίνεται. Ποια είναι η αντίθεση μεταξύ του τι θέλουμε και τι διατίθενται τα κράτη-μέλη να εισφέρουν. Γι' αυτό εξ αρχή είπαμε για του ίδιου πόρου τι θέλουμε. Δεν θέλουμε αυτό να είναι ο κύριο βασικό στόχο τη ε, πολιτική πρόταση που θα διαμορφώσει η Επιτροπή μα όσον αφορά τι ε, δημοσιονομικέ προοπτικέ. Όμω, οι ίδιοι πόροι θα αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα αυτή τη πρόταση που θα διατυπώσουμε. Και βεβαίω θέλουμε να υπάρχει ζωή περισσότερη Ευρώπη, να διατηρήσουμε όμω ε, τα, τα ίδια επίπεδα δαπανών και αυτό το οποίο μας απομένει είναι να διερευνήσουμε τους νέους πόρους που μπορούν να υπάρξουν για τον προπολογισμό. Βέβαια η διάθεση είναι πιο πολύπλοκη, δεν μιλούμε για απλή συγχρηματοδότηση, με τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει και το θέμα της προσθέμενης αξίας από τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Δεν είναι δηλαδή απλώς το 25% των διαρθρωτικών ε, ταμείων ή το 7% του Ταμείου Συνοχής έχει δική του προσθέμενη αξία ο, ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Έχει τους στόχους του που θα πρέπει να πετύχει. Είναι κάτι που πάει πέρα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και είναι κάτι που πάει πέρα από την συμπληρωματικότητα και την επικουρικότητα. Έχει του στόχου του κοινωνικού προπολογισμού και γι' αυτό η ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο και εργαλείο ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε προγράμματα κοινωτικά αποτελεσματικά. Ε, είναι ένα, ένα εργαλείο, ένα μέσο πολιτικής ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτές οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρόκειται να ε, συνεχιστούν και να δούμε τι θα γίνει με τις κοινωνικές πολιτικές και ε, ποιες από τις εθνικές πολιτικές θα ενισχύονται από τον κοινωτικό προϋπολογισμό. Ακούσαμε τις προάλλες στο Στασβούργο, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα πρακτικό έγγραφο το οποίο έχουν κατεβάσει και το οποίο βέβαια θα προκαλέσει αντιμαχόμενες απόψεις διότι τελικά το τι θα πει ε, ευρωπαϊκή προστέμενη αξία και αυτό είναι μια πολιτική κρίση για αξιολόγηση για την επίτευξη των πολιτικών στόχων. Για να δούμε δύο παραδείγματα. Πολιτική συνοχής, γεωργική πολιτική που είπε η κυρία Γκαρτιά Θάμπαλ ότι για μένα φυσικά και υπάρχει προσθέμενη αξία από αυτές τις πολιτικές. και έχουμε κάποιες μεθόδους ποσοτικής αποτίμησης, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργική πολιτική ούτως ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε πώς είναι η προσθεμένη αξία της ΚΑΠ, ας πούμε. Τι γίνεται με την ανάπτυξη της υπαίθρου, τι γίνεται με τις άμεσες ενισχύσεις. Δεν γίνεται. Έχουμε τη θέμενη αξία που δεν γίνεται να υπολογιστεί, να μετρηθεί ποσοτικά. Το ίδιο ισχύει για την πολιτική συνοχή και την ε, προστιθέμενη αξία που προσφέρει. Ή επίσης όσον αφορά την αναδυναμητική πολιτική ή τι γίνεται με κάποιους πόρους που έρχονται από κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιούνται για την ε, πολιτική αυτή και δημιουργούν ζήτηση, δημιουργούν ε, τζίρο σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτά πιστεύω και τα οποία τονίσαμε στην τελευταία μας συνάντηση. Έχω εδώ το κείμενο της κυρίας Χούμπνερ. Αναφέρει και κάποια χρήσιμα στοιχεία όσον αφορά ε, την ανάλυση της προστιθέμενης αξίας πριν την εκτέλεση των πολιτικών. Και προσπαθεί να ορίσει κάποιες παραμέτρους που καθορίζουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σύντομα θα έχετε και ένα κείμενο δικό μου όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος κατόπιν απόφαση των συντονιστών θα ξεκινήσει κάποια στιγμή ο δεύτερος γύρος προβληματισμού. Σας επαναλαμβάνω, ό,τι είπατε θα ληφθεί υπόψη για το εγγραφό μου. Και θεωρώ ήταν πολύ παραγωγική αυτή η συζήτηση και θα οδηγήσει σε ένα μεστό έγγραφο. Να δούμε τι θα γίνει με τις ε, επόμενες δημοσιογές πρόπτικες. Και μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση της στρατηγικής μας θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση και να συζητήσουμε τα της στρατηγικής εν του 2020. Ευχαριστώ όντως. Θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολλέ ε, σημαντικέ συζητήσει ακούσαμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θεωρώ ότι πλέον ο εισηγητή είναι σε θέση να καταρτήσει ένα έγγραφο το οποίο θα μα εκπροσωπεί όλου. Και τώρα περνάμε στο πέντε της ημερησίας διάταξης. Το δεύτερο θέμα. Θέλουμε να συζητήσουμε ποια θα είναι η στάση μας για τη στρατηγική του 2020 και σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί. Επικρατεί ασφαλώς ε, σχετική ομοφωνία. Έχει κάνει μια πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία και έχει εγκρίνει το Συμβούλιο και με μεγάλη πλειοψηφία έχει εγκριθεί και σχετικό ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει γενικά συμφωνία, υπάρχει κοινό τόπο. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να διαρθρώσουμε, να οργανώσουμε και να εντάξουμε αυτές, αυτούς τους στόχους και στον προπολογισμό. Και πάλι λοιπόν ε, κατήρτισε ένα έγγραφο ο Σάλβαντορ Γκαρίγκα το οποίο και θα αποτελέσει τη βάση της συζήτηση, συζήτησης. Όπως και προηγουμένως, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη ε, και τις εισηγήσει των συναδέλφων, θα καταρτήσουμε το έγγραφο εργασίας. Και εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω και τους δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ήρθαν εδώ σήμερα, ο Γενικός Διευθυντής κ. και ο Διευθυντής Λένα. Σας καλωσορίζουμε μετά την εισαγωγή του εισηγητή. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να λάβετε και εσείς το λόγο για να μας παρουσιάσετε τη σκέψη σας. Και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η δεύτερη φάση για τα οριζόντια θέματα όσον αφορά τη στρατηγική για το 2020 που θα είναι η γραμμή πλεύσης για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Και υπενθυμίζω εις όλους τους συναδέλφους ότι ο βασικός στόχος είναι να αποκτήσουμε κάποιες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013 αφού διαπιστωθεί το πόσο ολοκληρώθηκε η ζήτηση για τις προηγούμενες προοπτικές. Το να μπορέσουμε να αποκτήσουμε νέες τέτοιες δημοσιονομικές προοπτικές θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ένωση. Γιατί είχαμε μεγάλη διάσταση απόψεων. Και τα προγνωστικά ήταν ότι η συμφωνία θα επιτυγχανόταν δύσκολα. Και σας υπενθυμίζω ότι όταν συμφωνήθηκε την τελευταία φορά πια στην προοπτικές σοβούσε η χρηματοπιστωτική κρίση. Και πάλι θα έχουμε δυσκολίες 2011-2012 τα χρόνια που θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές συμφωνίες για τις προοπτικές. Θα είναι περίπλοκες διαπραγματεύσεις. Αυτές οι δημοσιονομικές προοπτικές χαρακτηρίζονται από συρρήκνωση της εισφοράς του κάθε κράτους μέλους. Αυτή θα είναι η αφετηρία για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και όπως είπε ο Πρόεδρος υπάρχει διοργανική πολιτική συμφωνία όσον αφορά τη στρατηγική του 2020 τοποθετήθηκε η Κομισιόν και το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο. Όπως συμφωνούμε με αυτή την στρατηγική για το 2020 και όπως μπορείτε να δείτε έχουμε τη σελίδα 2 του γράφου μελέτης για να διαπιστωθεί ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναδύονται τρία σενάρια ενώ του 2020. Πρώτα-πρώτα να φτάσουμε στο ρυθμό ανάπτυξης που έτρεχε το 2008 πριν αρχίσει η κρίση. Άλλο σενάριο, δεν θα υπάρξει ικανή ανάκαμψη. Να υπάρχει τόση ανεργία, τόσο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης που να γίνει το πρόβλημα διαρθρωτικό. Και υπάρχει και άλλο χειρότερο σενάριο να φτάσουμε στην κατάσταση της χαμένης δεκαετίας, 10-12 χρόνια δηλαδή που δεν θα υπάρχει ανάπτυξη, οπότε η κατάσταση θα είναι απελπιστική σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας του υπόλοιπου κόσμου. Οπότε, γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η στρατηγική του 2020, ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αποκτήσει την επιθυμητή ανάπτυξη. Ευφύ ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη. Φυσικά και το Κοινοβούλιο αναπαντώνει υπέρ αυτής της ιδέας και έτσι να έχουμε μια επιτυχή συνέχιση της στρατηγικής της Λισαβόνας. είχε γίνει ανάλυση της αποτυχίας της στρατηγικής. Είχαμε πει ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ πρικοδότησης και στόχων της πολιτικής αυτής. Όμως τώρα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία. Τώρα που καλούμεθα να χαράξουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές για να μπορέσουμε στην ίδια δέσμη μέτρων να συνδέσουμε επιτυχώς πολιτικές αποφάσεις με οικονομική χρηματοδότηση τα τρία θεσμικά όργανα έχουν συμφωνήσει ποιοι θα είναι οι στόχοι για την στρατηγική 2020. Επομένω, η συνέπεια είναι ότι οι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ θα πρέπει να είναι δομημένε, διαρθρωμένε επί τη βάση αυτή τη στρατηγική 2020. Αυτά θεωρητικά. Στην πράξη θα πρέπει να καταφέρουμε ο προπολογισμό να προσαρμοστεί στις μεταβολές των επιφέρουμε. Αλλά πάντως καταρχήν έτσι έχουν τα πράγματα. Και ελπίζουμε, ή μάλλον είμαστε σίγουροι, ότι η Κομισιόν θα ακολουθήσει τη δική μας γραμμή πλεύση. Αν κάποιος κάτσει και αναλύσει αυτή την πρώτη πρόταση σε την τη 2020 εκεί που έχουμε στη σελίδα 5 την πρόταση που κατέβηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον κύριο Λεβαντόφσκι και βλέπουμε τους βασικούς στόχους που αφορούν τα βασικά κονδύλια. Ε, Κάποιος μπορεί λοιπόν να εξετάσει τα σχετικά οικονομικά ποσά πρόκειται να εκπλαγεί βλέπουμε σε κάποιο τίτλο του προπολογισμού είναι 86% για αυτά τα flagships, αυτά το βασικό στόχους. Αλλού βλέπουμε ότι υπάρχει 25% σε σημαντική κατηγορία. Στην τέταρτη κατηγορία εκεί πάμε μόνο σε ένα 10%. Όλα αυτά τι σημαίνουν. Ότι η στρατηγική για το 2020 μέσω αυτών των flagships και το λέω στα αγγλικά γιατί μου φαίνεται ότι είναι πιο περιεκτική έννοια ενώ θα έπρεπε να κάτσουμε στη γλώσσα μας να αναλύσουμε περισσότερες λέξεις την ίδια έννοια επομένως πάμε σε ένα μόλις 3% των flagships σε σχέση με τον προπολογισμό για τη χρήση του 2011 και σας ερωτώ Τι έγινε με το υπόλοιπο 57%? πόσο πήγε ή τι, τι απέγινε αυτό που έπρεπε να πάει στην πολιτική συνοχή και την γεωργική πολιτική. Αυτό σας λέω για να σκεφτείτε. Σήμερα δεν μπορούμε να μετρήσουμε την δαπάνη στο βωμό της στρατηγικής 2020 γιατί αν θέλουμε να το κάνουμε θα πρέπει να εξαιρέσουμε πάρα πολύ ε, σημαντικά κονδύλια. Κάτι το οποίο φυσικά δεν το θέλει η Επιτροπή των Προπολογισμών. Για όλα αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δούμε τι γίνεται με όσο αφορά αυτά τα flagships. Πρόκειται για κάποιο μέσο κοινωνική πολιτική. Πρόκειται για προγράμματα. Πρόκειται για δεσμεύσεις πληρωμών και δαπανών. Πρόκειται για συνέχιση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πρόκειται για μεταβολή του τρόπου ορισμού, περιχαράκωσης κάποιων πραγμάτων σύμφωνα με το τι ζητάει ο κόσμος που εμείς από την πλευρά μας απλώς είναι ο Μανολιός που βάζει τα ρούχα του αλλιώς γιατί αυτό κάνουμε, ονομάζουμε τέτοια πράγματα με άλλα λόγια έτσι έγινε λοιπόν και γι' αυτό απέτυχε στα δική της Λισαβόνας έχουμε λοιπόν αυτό τον ωραίο καλοπισμό αυτό το μασκάρεμα για το flagship, για κάποιους βιώσιμους στόχους, αλλά όμως πίσω από αυτά δεν κρύβεται μια ξεκάθαρη δημοσιονομική πολιτική, άρα αυτό πάει προς βατερλό. Το κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να προσαρμόσει τις δημοσιονομικές προοπτικές σε αυτούς τους στόχους. Σήμερα πάντως δεν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις γιατί δεν έχουν οριστεί αυτοί οι βασικοί στόχοι, αυτές οι βασικές προτεραιότητες στα φλάξιψ αρκετά. Ξεκάθαρα. Βεβαίω και θα πρέπει να καλυφθεί η συνοχή και η γεωργία. Και υπάρχει εδώ πέρα μια όριστη υπόσχεση από πλευρά Συμβουλίου ότι δηλαδή η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχή πρέπει να στηριχτούν μέσω της συνήθιση της αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει επομένω, δεν, δεν αρκεί αυτό να λέμε έμεση υποστήριξη. Θα πρέπει για να, για να αυτέ οι πολιτικέ, θα πρέπει να αποτελούν ε, τμήμα του σώματο των, στόχων των πολιτικών τη στατική του 2020. Άρα η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, εξασφάλιση διατροφικής ασφάλειας, όλα αυτά φυσικά και είναι κριτήρια για την ΚΑΠ, κανείς δεν τα αμφισβητεί. Μιλάμε για πρώτο πυλώνα. Επομένως, ο πρώτος πυλώνας βεβαίως και θα πρέπει να καλύπτεται από τα flagships, από αυτές τις προτεραιότητες. Και αντίστοιχα, να καλύπτεται και από τι προβλεπόμενε δαπάνε τη αρχή 2020. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική συνοχή και το έχει πει πάνω κάτω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στην καρδιά αρχή 2020 είναι η κοινωνική εδαφική συνοχή. Βεβαίω, οπωσδήποτε αυτό και θα πρέπει να είναι κομμάτι της 2020, θα πρέπει να είναι μια δέσμευσή μας πάγια και συμφωνούμε ότι η πολιτική τη συνοχή θα πρέπει να αλλάξει ούτω ώστε να προσαρμοστεί, να ξεχρονιστεί, να γίνει πιο αποτελεσματική. Ίσως θα πρέπει να επανακαθαριστούν οι στόχοι της, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε στόχους με μέσα. Θέλουμε όμως μια πρώτη συγκεκριμένη της Κομισιόν για το πώς θα καλυφθεί η πολιτική της συνοχής από την πολιτική των δαπανών. Σας μεθυμίζουμε πάντως ότι υπάρχει εντολή του Κοινοβουλίου. Να υπάρχει επομένω καλά χρηματοδοτημένη ισχυρή πολιτική συνοχή που να καλύπτει όλη την Ευρώπη. Στα πλαίσια στεγής του 2020 επομένω είναι εντολή. Καλύπτει και τη δική μου εντολή και τέτοια πρώτα θα κατεβάσω. Ανακύπτουν τα διάφορα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να μας ενημερώσει σε σχέση με τις απόψεις της. Και συμφωνούμε ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την απόφαση επί των προοπτικών των δημοσιονομικών. Και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των flagships καλύτερα καθορισμένων σε σχέση με τις οικονομικές δεσμεύσεις της Κομισιόν και θα πρέπει να αντιστοιχούν αυτές οι flagships με τις κατηγορίες που προβλέπουν τις κατηγορίες δαπανών που προβλέπουν οι δημοσιονομικές προοπτικές. Επίσης, παρά το ότι δεν είναι τμήμα της ε, εντολής μας ως Επιτροπής, τι ευελιξία θα προσδοθεί σε αυτές τις flagships. Και σε σχέση με την γεωργική πολιτική, τι θα γίνει με την κατηγορία 4 των εξωτερικών δράσεων. Εδώ υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Γιατί μόλις το 10% καλύπτεται εδώ για τον προϋπισμό χρήσης 2000. Τι γίνεται με το πολύ 90%? Πώς θα το καλύψουμε? Γιατί η στατική 2020 θα πούμε ότι χρειάζεται λιγότερη εξωτερική δράση. Ανάλογα με την Ευρώπη που θέλουμε, ανάλογα με την προσθέμενη αξία που θέλουμε, πώς θα καλύψουμε την εξωτερική δράση. Έγινε με λεξιολογική διοτροπή που καθορίζει ότι πρέπει να είναι φλάξη η ιστορική δράση, αλλά βλέπουμε ότι το 90% ε, τη χρηματοδότηση που πρέπει να γίνει δεν καλύπτεται. Τι θα γίνει με τι διοικητικέ δαπάνε, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ανακύπτει. Επρόκειτο για βασικό θέμα συζήτηση στην Επιτροπή των Προπολογισμών. Επί πολλέ κοινοβουλευτικέ θητείε που τα ξέρει η πρόεδρο Χάουγκ δικέ δαπάνε θα μπορούσαν να πάνε όλε στην ίδια κατηγορία για λόγου αποτελεσματικότητα και διαφάνεια ή από την άλλη μεριά θα οι δικέ δαπάνε να τι κατανείμε σε διαφορετικέ κατηγορίε δαπανών. Εγώ θεωρώ ότι η πρώτη λύση είναι προτιμητέα. Επίσης, εδώ μιλούμε για τις προτεραιότητες. Εδώ βέβαια είναι θέμα πολιτικής απόφασης και άρα οι πολιτικέ ομάδε θα πρέπει να προγραμματιστούν και να αποφασίσουν ποιε θα πρέπει να είναι οι βασικέ προτεραιότητε για τι δαπάνε που θα ε, καλυφθούν από αυτέ τι ε, δημοσιονομικέ προοπτικέ. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί το τι προστιθέμενη αξία προέκυψε. Έχουμε και για αυτά τα περίφημα non-papers της Κομισιόν που προτείνουν ότι θα πρέπει στην έρευνα, στο διάστημα, στην ενέργεια, με μεταφορές, υποδομές να, να επικεντρωθούν αυτές οι προτεραιότητες, ε, παιδεία, νεολαία. Όλα αυτά είναι ε, θέμα προς πολιτική συζήτηση. Και σε σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. είπαμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν, το είπε και η πρόεδρος Χάουγ. Είχαμε συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και ενδιαφέρεται πάρα πολύ κυρίως το Πολεμικό Κοινοβούλιο γιατί προσεχώς θα αναλάβουν την Προεδρία της Ένωσης. Άρα θα εμπλαγούν και τα Εθνικά Κοινοβούλια σε αυτή την υπόθεση. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τα εθνικά προγράμματα όσον αφορά την στρατηγική του 2020. Επ' αυτού τα εθνικά κοινοβούλια έχουν πολύ σημαντικό έργο να επιτελέσουν. για το πώς θα συνδεθούν αυτά τα εθνικά προγράμματα με τη στρατηγική του 2020. Έτσι μόνο θα έχει σοβαρότητα η απόφαση για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Και όσον αφορά την ε, κατηγορία των δαπανών που είναι το τελευταίο τμήμα του, του εγγράφου Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στην επόμενη συνάντησή μα όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού, όσον αφορά τον τρόπο διαχείριση του κοινωτικού χρήματο. με γρηγόρησα λίγο, Πρόεδρε, αλλά έπρεπε να κάνω μια περίληψη αυτού του εγγράφου που είναι η εφετηρία προβληματισμού για τις πολιτικές ομάδες, για τους αδέλφους όλους αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί σε αυτέ μας τι ανησυχίε. Γιατί με λίγα λόγια δεν είναι δυνατόν ούτε η Επιτροπή μα ούτε ο υποφαινόμενο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ μια διαμόρφωση πρόταση για τι δημοσιονομικέ προοπτικές στα πλαίσια τη Στατική 2020 εάν δεν έχουμε επανακαθορισμό αυτών των flagships ούτω ώστε η κοινωτικέ δαπάνε να μπορέσουν να συντεριάξουν με την αντίληψή μα για στρατηγία το 2020. Σα ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο Ιούτα Χάουκ. Έχουμε, μπει έχουμε μάλλον συνηθίσει τι κάπως εκτεταμένε συνόψεις του εισηγητού μα. Θα παρακαλέσω ή δυνατόν να λάβει το λόγο η Κομισιόν. Αλλά πριν από αυτό θα σας διαβάσω ποιοι είναι στον κατάλογο γεγραμμένων. Danuta Hübner, Richard Ashworth Bas Es ist nicht das ähm, Es ist nicht das Ende der Δεν σημαίνει ότι κλείνει ο κατάλογος, αλλά για να ξέρετε ποιοι είναι γεγραμμένοι. Herr Generaldirektor. Σεις, κύριε Γενική Διευθυντά. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier. Euh, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή κύριο Καρίγα και για το έγγραφο που ε, υπέβαλε και για την ε, εκτεταμένη παρουσίαση. έθεσε μια ερώτηση πραγματικά μεγάλων διαστάσεων. Θα ήθελα να κάνω πρώτα κάποια σχόλια, σχετικά σύντομα. Και πρώτο, θυμίζω ότι η στατική του 2020 είναι ευρωπαϊκού επίπεδου. Δηλαδή, δηλαδή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Και σημαίνει μια δέσμευση κυρίως των χωρών μελών για την προσαρμογή των εθνικών πολιτικών για να επιτύχουν τον κοινά καθορισμένο στόχο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ορισμένα, ε, ορισμένοι μηχανισμοί, όπως γνωρίζει ο κύριος Γκαρίγα, έχουν ήδη ε, δημιουργηθεί. Η ευθύνη η κυρίως ευθύνη για την επιτυχία του 2020 λοιπόν ανήκει κυρίως στις χώρες μέλη και κυρίως οι χώρες μέλη είναι αυτές που πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να επιτύχει η πολιτική αυτή η οποία θα συνοδεύεται στο ευρωπαϊκό, στο κοινοτικό επίπεδο από τις δράσεις τις οποίες θα αναλαμβάνουμε εμείς κυρίως μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβλέψω τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεχώς ε, για την ενδιάμεση εξέταση του θέματος και τη σχετική ανακοίνωσή της που θα εκδοθεί στις 19 Οκτωβρίου. Μπορώ μόνο να πω, μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω προς τον κύριο Γκαρίγα ότι βεβαίως ο στόχος του 2020 βρίσκεται στο επίκεντρο των ε, προσπαθειών μας και των ανησυχιών μας και της αντίληψης συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία αντίληψη ε, επιθυμεί να θέσει στο κέντρο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου που θα συζητηθεί του χρόνου. Ουδεμία χωρί επί του προκειμένου αμφιβολία και θα ήθελα να πω επίσης ότι αναγνώσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα στοιχεία που διαλαμβάνει η έκθεσή του για την ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού στους στόχους 2020, για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, για την ποιότητα των δαπανών και για τις σχέσεις με τις Εθνικές Βουλές. Είναι σαφές ότι τα τέσσερα αυτά στοιχεία θα πρέπει να αποτελέσουν ε, το επίκεντρο της προσέγγισής μας. Υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις που τίθενται από πλευράς του κυρίου Γκαρίγα. Ασφαλώς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις απαντήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο της ε, ε, Επιτροπής σας. Εάν η στατική 2020 θα πρέπει να είναι η πολιτική αναφοράς για το μετά το 2013 για την Κομισιόν, στο ερώτημα αυτό απαντώ ναι. Πώς θα οργανωθούμε. Ο κ. Γκαρίγα θέτει ε, το πρόβλημα σε σχέση και με τους πίνακες που έχουμε διανύμει εδώ και λίγους μήνες για να δείξουμε ήδη με ποιον τρόπο ανταποκρίνεται ο κοινοτικός προπολογισμό στους στόχους 2020. Πώς θα οργανωθούμε λοιπόν. Αυτό είναι μια ερώτηση που θα απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δώσει κάποια στοιχεία απαντήσεων ήδη την επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά πάντα τις προτεραιότητες, συμφωνούμε με τον προβληματισμό που διαγράφει ο κ. Γκαρίγα και σε σχέση με το 2020 έχουμε το θέμα της συγκέντρωσης των δαπανών σε έναν αριθμό στόχων. Κάτι το οποίο θα μπει επίσης στο επίκεντρο των στοχασμών μας μέσα στην προοπτική της υποβολής των ε, απαντήσεων της Κομισιόν. Το πώς θα κατανεμηθούν οι στόχοι αυτοί στις διάφορες πολιτικές, πώς θα διαχειριστούμε τις πολιτικές, που θα πρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο ε, πλαίσιο, θα πρέπει να προσαρμόσουμε το πλαίσιο, θα πρέπει να προσαρμοστεί το πλαίσιο σε έναν αντικειμενικό στόχο ε, βέλτιστης αποδοτικότητας οι κατευθύνσει που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πολύ χρήσιμε για μα. Και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά είναι τα θέματα επί των οποίων τώρα εργαζόμαστε και μάλιστα με ιδιαίτερα ακριβή τρόπο. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των εθνικών προπολογισμών, είναι σημαντικό, νομίζουμε, και αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ε, προσέγγισης αυτής 2020, να διατηρηθεί το στοιχείο συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών δράσεων και των ε, δράσεων που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι, λοιπόν, οι διασυνδέσεις μάλλον με, τους, με τις εθνικές πολιτικές, με την ε, μορφή εξέτασης του τι συμβαίνει, είναι πράγματι ουσιώδες στοιχείο. Θα είναι πιο δύσκολο, πιθανόν, να φτάσουμε πραγματικά σε κάποια στοιχεία που θα μας επιτρέψουν στο επίπεδο της στατιστικής πλέον να κάνουμε συγκρίσεις ας πούμε επιστημονικού χαρακτήρα. Αν όμως μπορούμε ήδη να κάνουμε πρόοδους σε ό,τι αφορά την συμπληρωματικότητα και την ανάπτυξη αυτής της συμπληρωματικότητας νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό μέσα στα πλαίσια του επομένου δημοσιονομικού πλαισίου. Διεξήχθη συζήτηση πραγματικά θαυμάσια πριν από λίγο για την προστιθέμενη αξία και εμείς θεωρούμε ότι τίθενται ερωτήματα και για την ποιότητα των δαπανών και πρωτίστως της αιρεσιμότητας για τις δαπάνες στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Είναι και πιο γενικές ερωτήσεις σχετικά με την, αιρεσι, με την αιρεσιμότητα των δαπανών και την ανάπτυξη της οικονομικής διακυβέρνησης που επίσης ε, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων τις επόμενες εβδομάδες. Ιδού λοιπόν κυρία Πρόεδρε ορισμένα σχόλια που ήθελα να θέσω υπόψη σας. Νομίζω ότι και από το έγγραφο του κυρίου Γαρίγα και από την παρέμβασή του ε, ε, στην παρούσα συνεδρίαση διαπιστώνω σαφώς μια σύγκληση απόψεων για τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και αυτά που θα συζητηθούν στην επόμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα θέματα εκείνα που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να θέσει. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, κυρία Χάουκ. Ευχαριστώ. Α, εσείς Γιάννη. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα εδώ ο κύριος Μπέγκε, γιατί δυστυχώς ασθενεί και μου ζήτησε εξ ονόματος του να κάνω κάποια σχόλια. Η κυρία Πρόεδρος είχε πει ότι πλέον οι συντονιστές θα πρέπει να ε, μιλήσουν με διαφορετική σειρά. Αλλά εξ ονόματος του συντονιστή του ΕΛΚ θα ήθελα παρόλα αυτά να πάρω το λόγο σε αυτή τη φάση και να συμφωνήσω με όσα είπε ο εισηγητής μας, γιατί πολλά σημαντικά στοιχεία ανέφερε για την πολιτική του 2020, αλλά να επαναλάβω να αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όταν λάβαμε την απόφαση για τη στρατηγική της Λισαβόνας, τότε συμφωνήσαμε ότι η σημαντικότερη μέθοδος που θα έπρεπε να ακολουθηθεί ήταν η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού στην ευθύνη των κρατών μελών. Και τελικά προέκυψε και φάνηκε ότι δεν έτηρουν τις δεσμεύσεις τους ε, τα κράτη-μέλη. Τότε λοιπόν είχε ανακύψει το ερώτημα το πώς θα μπορούσαν οι άλλες ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν διαφορετική μέθοδο. Μιλήξαμε για την πολιτική συνοχή και πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί υπό το πρίσμα της στρατηγική τη Λισαβόνα και τελικά εφαρμόστηκε μόνο τμήμα της ε, πολιτικής συνοχής, δηλαδή η κοινωτική πολιτική τελικά χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και σήμερα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Ο εισηγητής μας εξήγησε το εξής. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, οι πολιτικές ε, οι οποίες ανέφερε, τις οποίες ανέφερε πριν από λίγο ο Γενικός Διευθυντής και ποια είναι η σχέση τους με τους ε, τίτλους του προπολογισμού. Αν το κάνουμε αυτό θα ξυνθούν τα προβλήματα και ύστερα έχουμε και τις ε, συμβατικές πολιτικές όταν τίθενται κάποιες ε, πολιτικές, κάποιοι στόχοι οι οποίοι δεν συνδέονται με κάποια στρατηγική αλλά αποτελούν αν θέλετε την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέτουμε λοιπόν κάποιους στόχους πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει σύνδεση και με τους στρατηγικούς στόχους από διοργανωτικής ε, πλευράς τώρα σε ό,τι αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούμε αλλά και σε ό,τι αφορά τους πόρους που χρησιμοποιούμε. Αν εξετάζουμε κατά πόσον οι πολιτικές εφαρμόζουν και βοηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων πέρα από τα χρήματα οικονομικά. Κατά πόσον ε, οι πολιτικές ε, βοηθούν την εκπλήρωση και περαιτέρω στόχων πέρα από την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Όλοι οι στόχοι λοιπόν, αυτοί που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για το 2020 αλλά και στις συνθήκες θα πρέπει να εξεταστούν. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος γιατί κατά το παρελθόν δεν υπήρξε ο σαφής αυτός διαχωρισμός των στόχων και αργότερα έπρεπε να προσαρμόσουμε τους στόχους στην πολιτική. Και σήμερα μας λέει ο εισηγητής ότι δεν είναι σαφές ότι η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική συμμετέχουν και βοηθούν στην επίτευξη των στόχων μας. Αυτό τι σημαίνει από πλευράς δημοσιονομικών. Σήμερα, για παράδειγμα, στην πολιτική συνοχής έχουμε το earmarking όπως ονομάζεται. Είναι πολύ σημαντικό μέσο ή ε, μήπω, θέλουμε να εφαρμόσουμε μια θεωρητική ιδέα. Θεωρώ ότι στη συζήτηση για το 2020 δεν μιλάμε θεωρητικά. Πρέπει να καθοριστεί αυτό η σύνδεση μεταξύ των στόχων που θα πρέπει να τεθούν και των λοιπών στόχων που δεν προκύπτουν μόνο από την στρατηγική για το 2020 και θεωρώ ότι δεν είναι σαφής ακόμα αυτή η σχέση επί του παρόντος. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος η κυρία Ντανούμπα Χίμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα τέσσερα σημεία να θίξω. Να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ε, αμφιβολίες μου για την στρατηγική του το 2020. Ωστόσο, αυτό για το οποίο δεν αμφιβάλλω είναι το εξής, ότι το η στρατηγική του το 2020 θα πρέπει να καταστεί ένα ευρωπαϊκό project βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά και να δώσουμε και μία όθηση στην ενότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι τόσο ιδιαίτερη η στρατηγική το 2020 για όλους μας. Και θα συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για μία κοινοτική, μία κοινοτική στρατηγική, αλλά εμείς ως Κοινοβούλιο θα επιμείνουμε στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλους τους τομείς, τους τομείς της στρατηγικής και ελπίζω επίσης στο σημείο αυτό ως κοινοβούλιο να επιδιώξουμε έναν ενεργό ρόλο του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, την εποπτεία της εφαρμογής των στόχων αυτών. Κατά δεύτερον, οποιαδήποτε στρατηγική για να είναι επιτυχής θα πρέπει να έχει μια ε, σύνδεση μεταξύ των στόχων και των μέσων των πολιτικών που έχει στη διάθεσή της. Άρα, για την Ευρώπη του 2020 σκεφτόμαστε και κοιτάμε ποια είναι τα πολιτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε τέσσερα σημαντικά μέσα, τα οποία έχουν έντονη διασύνδεση το ένα με το άλλο. Για τον ευρωπαϊκό, προ... προκειμένου ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να είναι αποδοτικός και να αξιοποιείται αποδοτικά, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ρυθμίσεις για την ιστορική αγορά που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής. Γιατί έτσι θα δοθεί νέα όθηση στην ανταγωνιστικότητα με την ανάλογη κοινωνική πτυχή και θα είναι πολύ πιο εύκολο με τον τρόπο αυτό να αξιοποιηθεί με αποδοτικό τρόπο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την εκπλήρωση και την ε, υλοποίηση της στρατηγικής Δεύτερο στοιχείο που σχετίζεται με τον ε, προϋπολογισμό είναι οι επενδύσεις κεφαλαίου που θα πρέπει να γίνουν σε όλες τις υποδομές, όχι μόνο στις μεταφορές αλλά και στις τηλεπικοινωνίες και το καθεξής. Και ξέρουμε ότι είναι τεράστιες οι ανάγκες και δεν μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά από εθνικούς και ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς. Χρειαζόμαστε διάφορους ε, συνδυασμούς, ε, διάφορες συνέργειες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και ενίσχυση των ε, χρηματοδοτικών οργανισμών της ε, Ένωσης. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συντονιστικός για την αξιοποίηση όλων των ε, μέσων. Τρίτος τομέας, οι εθνικοί προϋπολογισμοί αναφέρθηκαν. Στο σημείο αυτό να πω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει Σκοπός μας να είναι ο συντονισμός των εθνικών προϋπολογισμών, αλλά και ο συντονισμός των εθνικών προϋπολογισμών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και νομίζω ότι στους τομείς ε, προτεραιότητας της Ένωσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, η οποία μπορεί να βοηθήσει στα επόμενα βήματα. Και ένα νέο μέσο το Ευρωπαϊκό Μέσο Εξαμήνου. Θα πρέπει να υπάρχει η σχέση, η συμπληρωματική, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των Εθνικών και των Κοινωνικού Προϋπολογισμού, αλλά και περαιτέρω θα πρέπει να υπάρχουν και συνέργειες. Και έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, για τον οποίο θα είμαστε υπεύθυνοι. Νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της δικής μας Επιτροπής είναι ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών, αν θέλει, έχει την πολυτέλεια να εξετάσει κάθε αυτό τον προϋπολογισμό. Ενώ εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού και άλλων μέσων εφαρμογής της στρατηγικής. Άρα εμείς στην Επιτροπή μας θα πρέπει να εξετάσουμε τον προπολογισμό σε συνάρτηση με όλα τα υπόλοιπα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την επίτευξη και την υλοποίηση της στρατηγικής του 2020 και μιλώντας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θεωρώ ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η στρατηγική του 2020 δεν είναι τομεακής φύσης γιατί όλοι οι στόχοι που περιλαμβάνει είναι ουσιαστικά οριζόντια οριζόντιας διάταξης και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά το δυνατόν αυτή την ενοποιημένη προσέγγιση και θα πρέπει να συνδυάσουμε τα μέσα που έχουμε, τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να προωθήσουμε ένα άνοιγμα της στρατηγικής για να συμπεριλάβει και τον διεθνή ανταγωνισμό θα πρέπει να διοργανώσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να γεφυρώσουμε τα χάσματα που προκαλούνται από τις τομεακές προσεγγίσεις. Και τρίτον, να πω το εξής. Ε, παραπονιόμαστε συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν ε, ε, μαθαίνουμε από τα παθήματα της Λισαβόνας. Νομίζω ότι έχουμε αντλήσει πολλά διδάγματα και σε όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πολλά διαβάζουμε αναφορικά με το τι πήγε στραβά με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Και βλέπουμε σαφώς σήμερα ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν αρκεί να έχει καλούς στόχους, αλλά χρειάζεται και ένας μηχανισμός ε, ελέγχου των αποτελεσμάτων και ένας μηχανισμός εποπτείας. Και βλέπουμε επίσης με σαφήνεια ότι για τις ευρωπαϊκές πολιτικές χρειάζεται μεγαλύτερη εμπλοκή των ε, σχετικών φορέων και μεγαλύτερη εφαρμογή της επικουρικότητας καθώς και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Και τελευταίο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω, επειδή αναφέρθηκε η πολιτική συνοχή σε διάφορες περιστάσεις, να πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δύο-τρεις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτή της ε, ανακοίνωση που ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στο Λεξιμβούργο, τίθηκε το θέμα της ε, απόδοσης και σε ό,τι αφορά την στρατηγική της Λισαβόνας υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Άρα υπάρχει μια σωστή σύνδεση σε ό,τι αφορά την στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε την πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή αιρεσιμότητα και μια προσέγγιση βάσει των αποτελεσμάτων. Αν το πετύχουμε αυτό στη μεταρρύθμιση, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα και θα συμμετέχουν όλα τα επίπεδα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και ελπίζω ότι θα ανταπεξέλθει στις προκλήσεις η πολιτική συνοχής. και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν Γένσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Σαλβαδόρ για το εξαιρετικό έγγραφο προβληματισμού που και πάλι υπέβαλε που μας επιτρέπει να κάνουμε μια αναγωγή στις πηγές. Θέτει ορισμένα ερωτήματα εγώ θα προσπαθήσω να σας πω τις σκέψεις μου. Μία από τις σκέψεις που έκανε η ομάδα μου όταν διαβάσαμε το κείμενο, το έγγραφο, είναι αν θα συνεχίσουμε τα όσα ήδη έχουν κατατεθεί επιτάπητος. Ο κύριος Κάλφιν είπε ότι θα πρέπει να δεχθούμε ότι έχουμε περιορισμούς. Δεν μπορούμε να επανεφεύρουμε τον τροχό. Οφείλουμε να δεχθούμε ότι υπάρχουν κάποια κατεστημένα πράγματα και θα υπάρξει ίσως κάποια σταδιακή αλλαγή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την προοπτική να είμαστε και κάπως αδάμαστοι, ας πω έτσι. Ένα πράγμα που εμένα με κάνει να στοχαστώ ιδιαίτερα είναι στη σελίδα 6 του εγγράφου του Γκαρίγα όταν μιλεί για τίτλους και πώς να αντιμετωπίσουμε τη στρατηγική 2020 αν θα μπει στους τίτλους ή αν θα περιληφθεί στους τίτλους και η ερώτησή μου είναι γιατί έχουμε headings, τίτλους, γιατί αυτό δεν θα έπρεπε να συζητηθεί τον Νοέμβρη όταν θα συζητήσουμε την σύνταξη της δημοσιονομικής προοπτικής. Νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να αναρωτηθούμε, να συζητήσουμε γιατί στον προπολογισμό περιλαμβάνουμε τίτλους στα πολιετή προγράμματα. Αυτά είναι για να διευκολύνουν τις χώρες μέλη, γιατί όλες οι χώρες μέλη σκέφτονται αυτά που έλεγε τότε η Margaret Θάτσερ, δηλαδή θέλω τα λεφτά μου πίσω. Έχουμε όμως πολιετή προγράμματα, έχουμε μακροπρόθεσμα έργα, τα οποία πρέπει να χρηματοδοτούνται, να είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή τους δηλαδή. Ε, νομίζω, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν έχουν κάποιες, ε, κάποιο ενδιαφέρον οι, οι τίτλοι, γιατί πρέπει να στριμώξουμε μέσα σε τους τίτλους τις δαπάνες, ε, κάτι που νομίζω μειώνει την ευκαμψία του προϋπολογισμού. Τα είδαμε βέβαια αυτά και στην τελευταία δημοσιονομική προοπτική. Γιατί τίτλοι 3α, 3β που είναι πολύ μικροί περιγράφουν μικρούς τομείς οικονομικής πολιτικής, τα φτιάχνουν ένα είδος μικρό κοσμοδικό τους και μετά έχουμε ένα τεράστιο για την αγροτική ε, ε, οικονομία. Λοιπόν, πάντα σκεφτούμε αυτά. Επίσης, ε, κύριε Γκαρίγα, το, το ερώτημα εάν η στρατηγική του 2020 θα πρέπει να είναι το επικαλύπτων ας πούμε θέμα της επόμενης δημοσιονομικής προοπτικής. Εγώ ναι νομίζω θα πρέπει να είναι πολύ σημαντική αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν μπαίνουν στη στρατηγική 2020. Μιλήσατε για παράδειγμα για τις διοικητικές δαπάνες. Θα υπάρχουν και άλλα που έχουν σχέση με την διαχείριση, τη γενικότερη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως να μην μπορέσουμε να ταχώσουμε όλα στον τίτλο αυτό και νομίζω ότι δεν θα επακάνουμε καν την προσπάθεια. Νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχή, όπως είπε και η Ντανούτα Χούπνερ, θα πρέπει να εξετάζονται στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το κείμενο που λάβατε από το ψήφισμα για τη στρατηγική 2020, όπου ορισμένοι από εμά κάναμε σημαντική προσπάθεια για να πούμε ότι και η ε, αγροτική πολιτική πρέπει να μπει ως τμήμα της στρατηγικής. Γιατί αυτό που θα δούμε στο μέλλον είναι μια ε, δαπάνη ε, στην αγροτική οικονομία που θα έχει ως στόχο να διαμορφώσει μια σύγχρονη ανταγωνιστική γεωργία που θα προσφέρει βεβαίως ασφάλεια, προμήθεια τροφίμων, ποιότητα κλπ. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να στοχεύσουμε στην ανανέωση, στην καινοτομία στον τομέα αυτό. Και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε αυτό. Ε, ε, ρωτάτε ακόμα σχετικά με την συγχρηματοδότηση. Θέτεται δηλαδή το θέμα, ας πω καλύτερα, όπου νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής 2020 θα είναι σε τομείς που συγχρηματοδοτούνται. Όπως για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δείτε ότι ορισμένα έχουν μια τέτοια δομή που λέει ότι οι χώρες μέλη μπορούν να συμμετάσχουν και να χρηματοδοτήσουν ολόκληρο το έργο μόνες τους. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που προσφέρει είναι στην πραγματικότητα μια υποδομή τον τόπο συνάντησης, τους ιστοχώρους, τους κανόνες για το πώς να ε, λειτουργήσουν τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι πιο πλούσιες χώρες χρηματοδοτούν οι ίδιες ε, τη συμμετοχή των φοιτητών τους, τη συμμετοχή των ε, θεσμικών τους οργάνων και αλλού ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει την υποδομή χωρίς να χρειάζεται να χρηματοδοτήσει ολόκληρη την υπόθεση αυτή και ίσως οι ε, χώρες μέλη να χρηματοδοτούν κάπως περισσότερο από τώρα, από τη σήμερα. Τέλος, Λέτε να εξετάσουμε τα αποτελέσματα ή την απόδοση όταν εξετάζουμε τα προγράμματα και αν θα πρέπει να συνεχιστούν στο μέλλον. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών έχουμε το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο που έχει ως στόχο να μετακινήσει τις μεταφορές από ε, τις οδικές μεταφορές στις θαλάσσιες και στις ιδηροδρομικές. Είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο. Η Επιτροπή Μεταφορών είπε ότι ίσως πρέπει να επανεξετάσει αν χρειάζεται το πρόγραμμα αυτό ακόμη ή αν πρέπει τα χρήματα να διατεθούν αλλού. Αυτό έχει σχέση με την απόδοση, με, με, τα απόδοση αλλά και με τα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι προγράμματα τα οποία ήδη λειτουργούν κάποια χρόνια θα πρέπει να αξιολογηθούν, εάν θα πρέπει να συνεχιστούν ή όχι δηλαδή, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα νομίζω πρέπει να δεχτούμε ότι η Ένωση έχει λειτουργήσει ως καταλήτης, όπως για παράδειγμα στον τομέα της παιδείας. Και τότε όταν θα έχει παίξει τον καταλητικό ρόλο μπορεί να δεχθουμε οτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίσουν οι χώρες μέλη να χρηματοδοτούν. Αυτές λοιπόν είναι ορισμένες από τις ε, σκέψεις που κάναμε στην ομάδα μου πάνω στο έγγραφο χασμού σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σίγουρα είναι ενδιαφέροντα τα πράγματα αυτά και θα πρέπει να ε, καταβάλουμε προσπάθεια να καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ρίτσαρντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω τον Σαλβατόρο για την πολύ καλό έγγραφό του. Το διάβασα με πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Έχει συμπεριλάβει πολλές λεπτομέρειες και έχει θέσει πάρα πολλά ερωτήματα. Να πω όμως τέσσερα σημεία ήθελα να αναφέρω, Πρόεδρε. Το πρώτο είναι το εξή ότι οποιαδήποτε συζήτηση και αν γίνεται, πάντα καταλήγει στο μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και το στοιχείο αυτό θα ε, διατρέχει όλες μας τις συζητήσεις. Είναι θέμα πολιτικού οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ακούσαμε πολλές φορές σήμερα. Αν θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ ή πιο λίγη η Ευρώπη. Αυτό πάντα θα διατρέχει κάθε συζήτηση. Και εγώ συμφωνώ με την κυρία Πόλτσον η οποία ανέφερε ότι με τον περιορισμένο προϋπολογισμό θα πρέπει να αναζητήσουμε την αποδοτικότητα. Το more for less. Πιο πολλά με πιο λίγα. Προς το Σαλβαδόρ να πω το εξής. Έχουμε δύο βασικά τεστ για τις δαπάνες. Το θέμα της ε, επικουρικότητας ή το θέμα της αναλογικότητας. Και τώρα να κοιτάξουμε κατά πόσον προσθέτουν αξία και είναι η αξία αυτή ανάλογη των δαπανών. Δεύτερο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω. Συμφωνώ με τις ε, πιο πολλές απόψεις και τους πιο πολλούς στόχους που τίθενται στην στρατηγική του 2020 σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, ανταγωνιστικότητα, απασχολησιμότητα κτλ. Αλλά κάποια από τα στοιχεία αυτά επιτάσσονται από την ε, ανάγκη οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να διακρίνουμε δύο κατηγορίες. Καταρχάς, έχουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα, άμεσο όφελος, και εδώ αναφέρομαι όπως και η κυρία Χίμπνερ σε ε, επενδύσεις ε, στις μεταφορές, στις υποδομές, στις τηλεπικοινωνίες και του καθεξής και θα υπάρχει και ένα στοιχείο μακροπρόθεσμης, ε, μακροπρόθεσμου ωφέλους, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση, η διαβίου μάθηση. Και τα δύο είναι απαραίτητα, αλλά αυτό που μου προκαλεί σύγχυση είναι το εξή. Τα θέματα αυτά χάνονται κάπου στους γενικότερους τίτλους του προϋπολογισμού. Και καταλήγω στο τρίτο σημείο. Συμφωνώ με την κυρία Γένσεν. Δεν ε, θέλω να ενθαρρύνω τον ε, εισηγητή να θεωρήσει ότι δεν τον περιορίζει το ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Γιατί έχουμε την οικονομική κρίση επί του παρόντος και έχουμε τους όρους της συνθήκης της Λισαβόνας, είναι αξιοσημείωτη η ευκαιρία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν να καλέσω τον εισηγητή να επιδείξει φιλοδοξία και να αναπτύξει το όραμά του. Δεν ξέρω τι είπε η κυρία Γέντσα, νομίζω ότι είπε χρησιμοποιήσε τον όρο άγριο όραμα. Δεν ξέρω αν θα φτάσω μέχρι εκεί, αλλά εν περιπτώσει. Και τέταρτο σημείο. Πολλά ερωτήματα ερωτήματα τίθενται. Ίσως θα μπορούσε να διαμορφώσει ο εισηγητής ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε εμείς. Και έτσι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τα εθνικά κοινοβούλια στην συζήτηση αυτή. Να δώσουμε έναν κοινό χαρακτήρα, αν θέλετε, στις απαντήσεις που θα δοθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και πρωτού δώσω τον λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Έκχαουτ. Θα ήθελα να καλωσορίσω δύο πρώην συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύο πρώην βουλευτές, οι οποίοι θεωρώ ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το συνολικό Κοινοβούλιο αλλά και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή προϋπολογισμού. Όταν ξεκίνησα το 1994 εδώ, ο Τζον Κολόμπ ήταν ο κύριος δημοσιονομικές προοπτικές, να το πω έτσι. Και η Μπάρμπαρα Ντούρκοπ θα πρέπει να το πούμε ότι είναι, ότι η εφευρέ, είναι η εφευρέτρια των πλετικών ε, project. Υπό τη δική της ε, ηγεσία το ζητήσαμε αυτό από το Συμβούλιο. Τζον Κολόμπ και Μπάρμπαρα Ντούρκοπ, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Jetzt ist der <laughs> Der war's, ja. Äh. That's for you, äh, Mrs. Chairman. Thank you, thank you. Για, για σας το χειροκρότημα, Πρόεδρε. Σαλβαδόρ, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ αξιόλογο το έγγραφο της εισήγησης. Και πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η μέθοδος κάνει αυτό το αρχικό κείμενο, προβληματιζόμαστε και στη συνέχεια πάμε βαθύτερα. Πάρα πολύ καλή μέθοδος. Για να μην κινούμε εκτός θέματος. Και απέναντιλογούμε τώρα θα πρέπει να δούμε ότι και οι πράσινοι θέλουν το θέμα να προωθηθεί με κατεπήγοντα τρόπο, ίσως, ίσως να γίνει πιο άγριο. Ναι, ναι, διαλέγω προσεκτικά, Ρίτσαρντ τις διατυπώσεις μου να μην είναι τόσο ευγενική, τόσο μαλακή η συζήτηση απονευρωμένη γιατί θα καταντήσει κάτι θέμα ρουτίνας. Η πράσινη πάντοτε έχουμε επικρίνει αυτή τη στρατηγική του 2020 γιατί είναι σαν πολιτική κατευνασμού, είναι κάτι σαν ε, κάτι που τους βολεύει όλους. Τέλος πάντων, όλα τα άλλα θέματα θα πρέπει να καλύπτονται και για τον προπολογισμό επίσης. Είναι συρρικωμένος ο προπολογισμό σε σχέση με το σύνολο. Είναι προπολογισμό δαπανών. Πρέπει να ξοδέψουμε για να επενδύσουμε. Και αυτό έρχεται και δένεια με τη συζήτηση για την προσθέμενη αξία. Οπότε γι' αυτό και θα πρέπει να προετοιμαστεί για το μέλλον Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτόν τον άξονα πρέπει να προβληματιστούμε. Πόσο μα βοηθάει ο προπολογισμό να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Αυτό είναι το θέμα. Το κατεπήγον. Δεν είναι ακόμα μία κουβέντα σαν όλε τι άλλε. Είπαν οι συνάδελφοι, συμφωνούμε όλοι, μεγάλε οι προκλήσει. Όταν όμω έρχεται να χαράξουμε πολιτικέ τότε που καταλήγουμε στα γνωστά και πεπατημένα. Άρα, το θέμα κλειδί είναι κομμάτι της στρατηγικής για το 2020. Θα έχουμε σπάνιτα πόρων στο μέλλον και η οικονομία μας βασίζεται στη χρήση πόρων για απόκτηση πλούτου. Σε λίγο κόσμο έχει 9 δις 9 δις ή παραπάνω. Και αυτά τα 9 δισεκατομμύρια όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά για όλα τα πράγματα αντλούν τους πόρους. Γη, νερό. Εκεί θα δυσκολευτούμε εμείς και η Ευρώπη γενικότερα. Πώς δηλαδή θα αυξήσουμε τον πλούτο μας και ταυτόχρονα θα διαχειριστούμε αυτόν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους. Γι' αυτό και πρέπει να ρωτήμαστούμε. Και βέβαια σε κανένα δεν ε, αρέσουν τα παράπονά μας. Αλλά για κοιτάξτε καλύτερα. Τι γίνεται. Πανηγυρίζουμε για τους 33 μεταλλορίχους που απελευθερώθηκαν. Για κάτι να σκεφτείτε όμως γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, γιατί να πάνε εκεί. Ευτυχώς που σώθηκαν. Γιατί να βρίσκονται εκεί, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε την ολοένα και πιο επικίνδυνη άντληση πετρελαίου και εξόριξη. Όμως δεν είναι μόνο το θέμα η ενέργεια. Κίνα, Βραζιλία, χώρες τέτοιες δεν εμπορεύονται. Αγοράζουν γη για παραγωγή ενεργείας και ειδών διατροφής. Να, αυτό γίνεται σήμερα. Δεν τι έγινε με τα σιτηρά, την κρίση. Είχαμε αύξηση τιμή 40% πάλι. Να ποιο είναι το μέλλον. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως μπορεί να πει η Ευρώπη, περιμένουμε μέχρι ότι υπάρχουν αρκετά κίνητρα στις αγορές και να αναζητηθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι και χρήση. Ωραία. Α πούμε ότι συμφωνώ. Όμω από την άλλη μεριά μπορούμε να μια πολιτική απόφαση, να επιταχύνουμε περισσότερο τι εξελίξει και να διαλέξουμε εναλλακτικού τρόπου τώρα. Και αυτό για μένα έχει σημασία. Ότι όσο πιο πολύ περιμένουμε, τόσο το χειρότερο για την Ευρώπη. Γυράσκει ο πληθυσμό. Οι ρυθμοί ανάπτυξη δεν έχουν καμία σχέση με του ρυθμού Ινδία, Βραζιλία, Κίνα. Εμεί θα έχουμε ένα μισό εκατομμύριο πληθυσμό. Αυτή είναι πολλά δι. Μισό εκατομμύριο, αυτή πολλά δι. Επομένω, θα πρέπει να δούμε πώ με τι σωστέ αποφάσει δεν θα είναι αυτή πιο ισχυρή. Άρα θα πρέπει να επιταχύνουμε. Αλλιώς, αν περιμένουμε, θα μας περάσουν. Και μετά θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Να θεωρήσουμε ότι τα θέματα στρατηγικής του 2020 είναι κατεπήγοντα και το ίδιο είναι σχέση και τον προεπολισμό και τις δημοσιονομικές προοπτικές θέμα στο οποίο περνώ τώρα. Ναι. Θα πρέπει ο όντω να λεμπορήσει δικτυοκαλλιέργειες είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα ένταση σπόρων τομέα. να η πρόκληση άρα η θα πρέπει να δει τώρα πως θα μπορέσει να διατηρήσει στα επιθυμητά επίπεδα την παραγωγή αλλά με χρήση γίνεται λιγότερων πόρων και έτσι η ηχθειοκαλλιέργεια να γίνει κλειδί επιτυχίας για το μέλλον. Επομένω, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Το ίδιο ισχύει για τι πολιτικέ αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί. Για να προετοιμαστούμε για το μέλλον, για να αναδιαθρώσουμε την οικονομία μα, για να έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, τότε κάποιοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητα θα βγουν χαμένοι καταρχήν. Θα πρέπει να υπάρξουν θυσίες σε κάποιους κλάδους, σε κάποιες περιοχές. Και για αυτό και χρειάζονται πολιτικές συνοχές για να βοηθήσουν. Και τις υποδομές, ενεργειακές υποδομές επίσης, θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Να γίνουν επενδύσεις έρευνα και ανάπτυξη. Τώρα γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν επενδύουμε αρκετά, δεν υπάρχει κατανομή άνηση, εξωτερικές πολιτικές επίσης, γεωπολιτικά, θα πρέπει να τα σκεφτούμε καλύτερα. Και ελπίζω ότι σας πείθω ότι πρόκειται για κάτι που επήγε. Πολύ σημαντικό το είπε ο Σαλβαδόρ για το αν χρειάζεται η ιδιωτικοποίηση. Ναι, λέω εγώ. Η στρατηγική η 2020 είναι πάρα πολύ βασική, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Θα πρέπει τα σημαντικά θέματα να τα αναδείξουμε, Ρίτσαρντ, να είμαστε πιο φιλόδοξοι και έτσι να έχουμε ιδέες πρωτότυπες και δεν σας θέλω αυτά σαν ρομαντικός. Δεν ονειροπολώ. Σύμφωνοι, μπορούμε να πούμε καθόμαστε τα χέρια σταυρωμένα μέχρι ότου η αγορά βρει τη λύση. Ωραία, εγώ όμω λέω θα είναι πολύ καλύτερο εάν από τώρα φροντίσουμε. Αν προχωρήσουμε με τέτοιο ζήλο και ορμή όπως ε, ε, μόλις τώρα ο Μπάς, τότε σίγουρα θα ε, έχουμε μεγάλη επιτυχία. Βέβαια δεν θα πούν όλοι τα ίδια. Α, αυτοί οι πράσινοι και οι σπάνιοι των πόρων την οποία επικαλούνται. Έχουμε τώρα και άλλα πράγματα να ακούσουμε. Γιατί και ο σύνδεσμος γερμανικών βιομηχανιών μιλούν ε, για, ε, μιλεί για ε, σπάνιδα πόρων και βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι μέλη των πράσινων. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, πολλές άλλες πτυχές. Η κυρία Γκόνς δεν ξέρω αν και εγώ θα μπορέσω να συνεχίσω με την ίδια ορμή, αλλά πιστεύω από τη μια μεριά ότι κινδυνεύουμε να κάνουμε δύο λάθη και ίσως προσπαθήσουμε να βρούμε ένα ενδιάμεσο δρόμο. Ένα λάθος θα μπορούσε να είναι να προσπαθήσουμε δηλαδή να επιδιώξουμε μηχανικά τη στατική 2020 και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις επικεφαλίδες του προπολογισμού ένα προς ένα. Γνωρίζουμε ότι η στρατηγική 2020 επιθυμεί ένα διαφορετικό τρόπο, επιθυμεί να θεσπίσει ένα διαφορετικό τρόπο εφαρμογής. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πέρασμα ε, στους τίτλους του προπολογισμού δεν θα είναι εύκολο. Λοιπόν, όπως είπα, το ένα λάθος θα μπορούσε να είναι αυτό. Και να αφήσουμε εκτός άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στη στρατηγική 2020. Άλλο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι εάν δεν ε, λάβουμε υπόψη επαρκώς τη στρατηγική αυτή στην έγκριση του προπολογισμού. Άρα, όπως είπα, ανάμεσα στα δύο άκρα καλό είναι να βρούμε ένα μέσο, μια μέση οδό. Ο πίνακα τη σελίδα 5 ε, είναι εντυπωσιακό, Μιλώ δηλαδή για τις ε, βασικές εκείνες πρωτοβουλίες, τις flagship initiatives και τους σχετικούς πόρους. Δύσκολα μπορούν να εκφραστούν αυτά ε, βέβαια με αριθμούς όπως ε, για παράδειγμα οι στόχοι των ε, τίτλων. Επίσης οι πόροι για την καινοτομία για παράδειγμα εύκολα μπορούν να διατυπωθούν με αριθμούς. Όταν όμως μιλούμε για απασχόληση για παράδειγμα το θέμα εκεί είναι πολύ πιο περίπλοκο. Αν όταν καθίσουμε να μιλήσουμε μαζί για ε, πολιτική αναβληση πέθρου, για κοινή αγροτική πολιτική, θα δούμε ότι εκεί παίζουν σημαντικό ρόλο πολλοί παράγοντες. Θα ήθελα λοιπόν <clears throat> να σας ε, επιστήσω την προσοχή ότι δεν πρέπει να ε, είναι μηχανικός ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, δηλαδή ένα προς ένα με τον προϋπολογισμό. Επίσης οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να έχουν υπόψη τους στη στατική 2020 και εν προκειμένου το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι καλός τρόπος προσέγγισης κυρίως ό,τι αφορά την διαφάνεια. Θα δούμε δηλαδή τι γίνεται στην φάση σχεδιασμού του προϋπολογισμού και ίσως μπορούμε να την επηρεάσουμε. Άλλο ε, θέμα, εάν θεωρούμε σωστούς και σημαντικούς τους στόχους της στρατηγικής, πρέπει να δούμε και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση. Άρα θα υπάρξουν στόχοι που θα πρέπει να επιτύχουμε προηγουμένως, καθήκοντα που θα πρέπει να, επιτύχουμε, να, ασκήσουμε προηγουμένως και άλλα που θα χρειαστεί να αναβληθούν και ε, σε ό,τι αφορά τους πόρους. Επίσης, άκουσα πολλά για φυσικούς πόρους. Εγώ θα αναφερθώ στις δαπάνες που έχουν σχέση με τους ανθρώπινους πόρους, που είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικοί με τους φυσικούς. Είναι σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε ε, ποιε είναι οι πηγέ των πόρων αυτών. Ναι, μάλιστα πρέπει να διασυνδεθούν αυτά τα πράγματα. Όταν μιλούμε για αποδοτικότητα τη ενέργειας, για ε, εξοικονόμηση πόρων, Πρέπει τότε να μιλήσουμε και για παιδεία, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση, οτιδήποτε θέλετε. Όλα αυτά δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. ΕΙΔΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι περισσότεροι και περισσότερες από μας είναι είμαστε οπαδοί της στρατηγικής 2020. Και στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που οδήγησαν στην αποτυχία της στρατηγικής Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα γιατί δεν θα μας το συγχωρήσει το κοινό Πρέπει να φροντίσουμε να επιτύχει η στρατηγική του 2020. Επίσης είναι σημαντικό να φροντίσουμε ώστε η στρατηγική αυτή να σέβεται τους περιορισμούς του προϋπολογισμού, όχι όμως μόνο αυτό. Θα υπάρξουν ορισμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα 3α, 3β, 4, που θα ενταχθούν στη στρατηγική 2020 και άλλοι που δεν θα ε, ενταχθούν σε αυτήν. Άλλες όπως ε, η στρατηγική της κοινή αγροτικής πολιτικής πρέπει να θεσπίσει στόχους που θα μπορέσουν να επιτευχθούν αλλά δεν θα μπουν όλα τα πράγματα μέσα στη στρατηγική του 2020. Φοβούμε μήπως ξεχάσουμε ορισμένα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει διαρκώς. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα ότι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και να ε, ρηχτούμε μόνο σε αυτή τη στρατηγική του 2020. Βεβαίως θα βασιστούμε στο παρελθόν και θα προχωρούμε με καινοτόμο σκέψη προς το μέλλον. Όμως δεν μπορούν όλοι οι στόχοι να είναι αποκλειστικά η χρηματοδότηση της στατικής του 2020. Στο έγγραφο διαλαμβάνονται πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα και ποιος θα είναι ο ρόλος των χωρών μελών και των εθνικών προϋπολογισμών. Αλλά μη λησμονούμε ότι ο προπολογισμό μας δεν είναι παρά το 1% του συνολικού προϊόντος των ε, χωρών μελών. Άρα θα χρειαστεί να ε, εγγύψουν και αυτές ε, στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που οι χώρες μέλη θα είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές για να λειτουργήσει η στρατηγική αυτή και ελπίζω να δεσμευτούν γιατί αυτό υπήρξε και το σφάλμα που κάναμε στην ε, στρατηγική της Λισαβόνας που δεν δεσμεύτηκαν οι χώρες μέλη δηλαδή για την ε, υλοποίησή της. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις ακόμα που θέτει ο ε, Σαλβαδόρ Γκαρίγα. Χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για να οριστούν καλύτερα αυτά τα πράγματα, αλλά προς Θεού ας μην χάσουμε άλλη μια τέτοια ευκαιρία, γιατί αυτό θα σημαίνει καταστροφή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ακούστε πάλι τα ονόματα. Jürgen Klute, Herr Sikierski, äh, De Jong und ähm, Ivalo Kalfin. Und dann bindet äh, Salvador ab. Και μετά θα ολοκληρώσει και θα μας μιλήσει ο κύριος Γκαρίγκα. Ευχαριστώ, Γιούτα. Το ακούσαμε και στην αρχή ότι η στρατηγική για το 2020 ε, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στο Κοινοβούλιο. Να πω όμως ότι η ΓΚΟΕ, η ομάδα μου, έχει μια πιο επιφυλακτική και κριτική στάση σημειώνουμε ότι σε αντίθεση με τη στρατηγική της Λισαβόνας η θεματική βασίζεται στον κοινωνικό, στο κοινωνική πτυχή και αυτό το καλωσορίζουμε ασφαλώς, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η στρατηγική για το 2020 συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο την πολιτική για τον ανταγωνισμό που είχε ξεκινήσει η στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία και οδήγησε σε ανισότητες στην Ευρωζώνη, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα το κατά πόσο ο στόχος αυτός της εντονότερης ε, κοινωνικής συνοχής μπορεί να επιτευχθεί με παράλληλη συνέχιση της πολιτικής ανταγωνισμού που είναι αντίθετη πέρα από το κατά πόσο ο προπολογισμό αρκεί για να επιτευχθούν τα ελλείμματα, να επιτευχθεί η πλήρωση των κενών που υπάρχουν. Μια δεύτερη πτυχή. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μιλάμε αφηρημένα για στόχους και το κάνουμε και πρέπει φυσικά να το κάνουμε γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε το τι μας απασχολεί πολιτικά αλλά να κοιτάξουμε και τι συμβαίνει επιτόπου, γιατί προέρχομαι από μια περιοχή ε, η οποία έχει λάβει πολλά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις υποδομές και αυτό φυσικά ξέρω ότι έχει και μία πιο επικριτική ε, πτυχή αλλά πολλά θετικά έχουν επιτευχθεί αν ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε στόχους σε, σε αφηρημένο επίπεδο θα πρέπει να κοιτάξουμε τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί επί τόπου στις περιφέρειες έχουν συμβεί μόνο αρνητικά πράγματα ή μήπως υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Υπάρχουν θετικά στοιχεία πιστεύω και αν θέλουμε να σταματήσουμε κάποια προγράμματα ενίσχυσης, αν θέλουμε να συνεχίσουμε κάποια άλλα μέσα, αυτό δεν είναι αντικείμενο κριτικής, απλά να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες του να σταματήσουμε για παράδειγμα κάποια προγράμματα. Να προσέξουμε λοιπόν ποια θα είναι η στοχοθέτησή μας για να μην απέχει πάρα πολύ αυτή η στοχοθέτηση από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γιατί πολύ συχνά υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρυνόμαστε από την πραγματικότητα, από τον πολίτη. Δεν είναι φυσικά σωστό αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαμεσολαβούμε εξ ονόματος των πολιτών. Άρα, να κάτσουμε και να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί με τα κονδύλια ως τώρα και κατά πόσο αξίζουν όλα τα προγράμματα να συνεχιστούν. Δεν μπορούμε δηλαδή να, τα αντικαταστήσουμε όλα. Να δούμε μήπως κάποια από τα προγράμματα αξίζει να συνεχιστούν. Και το είχε αναφέρει και ο κύριος Άλβαρο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την προστασία προστασία και εκτιμένη σε κάποιες περιπτώσεις αξίζει να διατηρηθούν κάποια προγράμματα Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή ο κ. Σικιάσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητήσαμε τις τεχνικές πτυχές αναφορικά με τον συντονισμό των συνεδριάσεών μας ε, με τις άλλες επιτροπές. Ε, Νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να απαντήσουμε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν και το παρόν, αν θέλετε, της πολιτική μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση έχει ω εξή. Μπορεί κάποιες χώρες να έχουν αντλήσει τα διδάγματα από την κρίση. Δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουμε χρησιμοποιήσει τα λάθος ε, μέσα μπορεί να μην έχει εφαρμοστεί οι διατάξει του Συμφώνου Σταθερότητα. Αλλά πού ήταν ο Ευρωπαϊκό Έλεγχο, πού ήταν τα ευρωπαϊκά μέσα όταν τα χρειαστήκαμε, γιατί καταλήξαμε στην κατάσταση αυτή. Έχουμε ελέγχου αναφορικά με τα αποτελέσματα, οι οποίοι όμω δεν ε, ήταν επαρκεί τελικά. Και από αυτό προκύπτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την κρίση. Αναφορικά με το μέλλον λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν συζητούμε λοιπόν στην Επιτροπή, στη δική μας Επιτροπή για το μέλλον, να αναρωτηθούμε κατά πόσον θέλουμε να αλλάξουμε κάποια στοιχεία και κατά πόσον κάποιες άλλες πτυχές θέλουμε να παραμείνουν απαράλλαχτες. Γιατί δεν βλέπουμε ποιε ήταν οι επιτυχίες, για παράδειγμα, στην πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής προκάλεσε τις εξελίξεις, για παράδειγμα, στον τομέα της επιστηστικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα να επιδείξουμε, θεωρώ. να προσαρμόσουμε για παράδειγμα την αγροτική πολιτική, την πολιτική συνοχής, όπως προβλέπεται στις συνθήκες σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του του άνθρακα, σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θεωρώ ότι η στρατηγική το 2020 δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στις προσδοκίες μας, αλλά αυτό δεν ήταν το ζητούμενο απαραίτητα. Να σκεφτούμε πώς προέκυψε άλλωστε η στρατηγική αυτή. Θεωρώ ότι οι εργασίες της Επιτροπής μας θα δώσουν, αν θέλετε, ζωή στην στρατηγική αυτή και αναμένουμε και σημαντικά έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βιαστεί και να μας υποβάλει τα έγγραφα αυτά που περιμένουμε. Μέχρι το 2014 έχει ακόμα τρία χρόνια στην διάθεσή της. Μέχρι το 2020 έχουμε, ε, ας πούμε, 10 χρόνια ακόμα. Και ως προς την ευελιξία, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, η ευελιξία μας για αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς ε, θέλουμε, για παράδειγμα, να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει ήδη από σήμερα να κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Και νομίζω ότι κάνουμε μια σωστή αρχή, αν θέλετε, στο σημείο αυτό στην Επιτροπή μας συζητάμε κάπως γενικά για το παρελθόν, χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς συγκεκριμένα μέτρα, αλλά να εξετάσουμε και αυτά που πήγαν στραβά στην στρατηγική της Λισαβόνας. Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, για παράδειγμα, και πώς διαμορφώθηκε. Και τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ για τις πολιτικές αυτές. Απλά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσοστό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος Διγιώμ. Είναι εξαιρετικό το reflection paper ε, του συναδέλφου και να τον ευχαριστήσω, αλλά θα ήθελα να αναφέρω τρία θέματα. Καταρχάς, το πόσο είναι μετρήσιμη είναι και πόσο ε, δημοφιλής είναι η πολιτική. Εγώ από την αρχή προσπαθώ να εκπροσωπήσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μίλησα ήδη χθε με πολλού από αυτού. Ένα βασικό θέμα το οποίο απασχολεί κάθε επιχειρηματία είναι το εξή. Ωραία είναι τα λόγια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μα λένε, αλλά πώ μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αν το κοιτάξουμε αυτό αναφορικά με την στρατηγική το 2020, όντως πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ ασαφείς ε, και αφηρημένες ε, οι έννοιες που αναφέρονται. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να επιτευχθούν το συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη στοχοθέτηση για την καταπολέμηση της ένδυας, την απασχόληση, σημαντικά θέματα, αλλά με πολύ αφηρημένη διατύπωση. Νομίζω λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι μια χαρά, αλλά θέλουμε πλέον πιο συγκεκριμένα χαρακτήρα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά την, ε, τους πόρους. Μία συνέντευξη τύπου της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών ε, αναφέρθηκε ότι θέλουμε πιο πολλούς πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι πολύ λάθος ο τρόπος αυτός για την παρουσίαση της Ευρώπης στο κοινό. Κάθε εθνική κυβέρνηση δηλαδή ε, παίρνει μέτρα λιτότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βγαίνει και να ζητάει πιο, πολύ χρήματα, πιο πολλά χρήματα. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό. Πρέπει να υπάρξουν ε, οικονομίες και να δούμε με κριτικό τρόπο τους πόρους που διαθέτουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντανακλαστικά ζητούν τα κράτη-μέλη πολλά ταμεία χρηματοδότηση και προκαλούνται έτσι μεγάλος βαθμός ε, χρηματοδότησης και πολλά επίπεδα Τη Ευρωπαϊκή πολιτική δεν αξιοποιούνται και αυτό είναι κρίμα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα ήταν υγιέ να εξετάσουμε εκ νέου τα ταμεία αυτά, του σπόρου αυτού με δύο τρόπου. Καταρχά, θα πρέπει ασφαλώ να είμαστε αλληλέγγυοι στην Ευρώπη, γιατί ήρθαν και προσθέθηκαν χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι, οι οποίοι συστερούν και θα πρέπει λοιπόν ένα ε, τμήμα των κονδυλίων να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις χώρες. Και κατά δεύτερον, να κοιτάξουμε τι χρειάζεται η Ευρώπη για το μέλλον. Και όντω χρειαζόμαστε βιωσιμότητα και γνώση και καινοτομία και φυσικά θέσεις απασχόλησης. Αν προσανατολιστούμε σε όλα αυτά και θέσουμε τα κριτήρια αυτά για την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης, ζητήσουμε διασυνοριακά project και επίσης να λάβουμε υπόψη ότι θα υπάρξει μια συγκέντρωση σε ό,τι αφορά την καινοτομία Θεωρώ λοιπόν ότι στους τομείς αυτούς θα έπρεπε να αξιοποιηθούν οι πόροι σε ό,τι αφορά και την στρατηγική του 2020. Κάτι τελευταίο για τις εθνικούς προϋπολογισμούς. Μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί είναι συμπληρωματικοί με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Με κάθε σεβασμό και αν δεν κάνω λάθος θεωρώ ότι ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός είναι συμπληρωματικός προς τους εθνικούς. Αυτό πρέπει, θα, είναι, θα πρέπει να είναι το σημείο αφετηρίας. Δεν θα πρέπει να αγοράζουμε, να προσπαθήσουμε να αγοράσουμε, αν θέλετε, να εξαγοράσουμε τα κράτη-μέλη μέσω των κονδυλίων. Όχι, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές συμφωνίες. Και το βλέπουμε αυτό σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική πειθαρχία. Τίθεται το θέμα των κυρώσεων. Αυτό δεν ε, υπάρχει, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στοχοθετήσεις στην πολιτική τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020. Το συζήτησα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να μην έχουμε έτσι πιο αυστηρό καθεστώς σε ό,τι αφορά τους πόρους για την καταπολέμηση της έντιας για παράδειγμα. Θα πρέπει να υπάρχει η ίδια πολιτική δεσμευτικός, ίδιος πολιτικός δεσμευτικός χαρακτήρας και επίσης να ελέγξουμε και να ελέγχουμε διαρκώς την αποδοτικότητα όχι μόνο την νομιμότητα των δαπανών, αλλά και την αποτελεσματικότητά τους, προκειμένου να είναι πιο αξιόπιστη η Ευρώπη χωρίς επιπλέον κόστος. Σας ευχαριστώ, Κάλφιν. Ευχαριστώ. Το έγγραφο προβληματισμού του Σαλβαδόρ όντως μου προκάλεσε πολλές σκέψεις και για το λόγο αυτό αποδεικνύει την αξία του. Προκάλεσε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ. Εγώ νομίζω ότι είναι και ευτυχής η σύμπτωση ή ας μην πω σύμπτωση καλύτερα, αλλά αρχίζουμε και συζητούμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και προχωρούμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο μετά, που είναι η Ευρώπη του 2020 γιατί, γιατί η προστέμενη αξία είναι πολύ γενική συζήτηση. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς του προϋπολογισμού για να επιτύχουμε κάποια προσθέμενη αξία. Εγώ συμφωνώ ότι η Ευρώπη του 2020 αποτελεί προτεραιότητα που δεν μπορεί να αναφέρεται σε όλα τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συμφωνώ με τον Γενικό Διευθυντή που είπε ότι είναι συνολική ε, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο των θεσμικών οργάνων, αλλά και των χωρών μελών. Αυτό που θα χρειαστεί να δούμε είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο του προϋπολογισμού για να επιτύχουμε αυτούς τους ευρύς πολιτικούς στόχους. Εδώ τίθεται το θέμα πόσο μπορεί να συμβάλλει ο κοινοτικός προϋπολογισμός, σε ποιο βαθμό, τι μπορούμε να αναμένουμε από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεύτερο, τι είδους έργα μπορεί να χρηματοδοτήσει. Έχουμε τις flagship initiatives. Έξοχα. Η ιδέα υποθέτω ότι είναι να αποτελέσουν μια μηχανή έλξης των προτεραιοτήτων αυτών που θα χρηματοδοτηθούν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και αναφανεί ότι υπάρχει, σημειώνεται μια σαφής πρόοδος. Μιλούμε επίσης πολύ σήμερα εδώ για αποδοτικότητα, που δεν μπορεί κανείς να τη μετρήσει όμως αν δεν έχει στόχους. Άρα έχουμε τις flagship initiatives, δεν ξέρουμε όμως τι ακριβώς θέλουμε. Ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, ξέρουμε ποιες είναι οι σημαντικές πολιτικές, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε μέχρι το 2020. Αν τα ξέρουμε αυτά, τότε μπορούμε να πούμε εάν είναι αποδοτικό ή όχι να χρηματοδοτηθούν από, ευρωπαϊκά, από ευρωπαϊκούς πόρους. Οι πρώτες ερωτήσεις είναι σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να επιτευχθούν συνολικά αυτές οι προτεραιότητες. Το δεύτερο έχει πιο ουσιώδη χαρακτήρα. Έχουμε ορισμένους στόχους. Στην Ευρώπη 2020 έχουμε μάλιστα σαφείς στόχους για το τι θα πρέπει να επιτύχει η Ένωση μέχρι το 2020. Έχουμε τρεις τρόπους χρηματοδότησης και μιλώ μόνο για τους χρηματοδοτικούς πόρους και όχι για άλλους τρόπους που ίσως να μην συνεπάγονται χρηματοδότηση. Πρώτα, τα νέα ευρωπαϊκά ταμεία. Είτε λοιπόν απολύτως νέα, είτε αναδιάρθρωση η οποία να διαθέσει εξοχήν, κατά πρώτον λόγο δηλαδή, ορισμένα ε, κονδύλια σε ορισμένα ε, ταμεία. Δεύτερο, το earmarking. Συμφωνώ την άποψη του Γαρίγα για τη δήλωση της Επιτροπής ότι 43% του κοινοτικού προϋπολογισμού ήδη κατευθύνεται σε στόχους του 2020. Άρα λοιπόν ή δεν αλλάζουμε τίποτα, είτε κάνουμε κάποια αναδιάρθρωση σε κάποιες προτεραιότητες και με τον ίδιο προϋπολογισμό, όπως και να τον αποκαλέσουμε, προχωρούμε. Αυτά νομίζω είπε περίπου και ο Σαλβαδόρ. Τέλος πάντων, έχουμε αυτό το μηχανισμό, το earmarking των ε, υφισταμένων προγραμμάτων και ποιο τμήμα από αυτά μπορεί να δοθεί για τους στόχους 2020. Έχουμε και άλλες ε, ε, πηγές, πηγές χρηματοδότησης που είναι οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Είτε συγχρηματοδοτώντας, είτε με δικά τους εθνικά κονδύλια και προτεραιότητες. Με τους εθνικούς προϋπολογισμούς έχουμε δύο προβλήματα Πολύ σημαντική βέβαια, χρειάζεται συντονισμό μαζί του, αλλά τι ακριβώ πρέπει να συντονίσουμε. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι πολλέ χώρε μέλη και έχουμε και την εμπειρία τη στρατηγική τη Λισαβόνα, πολλέ λοιπόν χώρε μέλη δεν ανταποκρίνονται στου στόχου αυτού. Για παράδειγμα, το 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και ανάπτυξη. Πολλέ πολλές χώρε δεν ε, υλοποίησαν το στόχο αυτό. Θα ήταν ίσως μια ιδέα. Θα συζητήσουμε βέβαια και την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Όπως όπου έχουμε στόχους που έχουν εγκρίνει οι χώρες θα πρέπει να ε, είναι πιο δεσμευτικοί οι στόχοι. Όπως γνωρίζετε τα έχουν αναλάβει μόνες τους οι χώρες αυτές εθελοντικά. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε διαφορετική ικανότητα των ε, εθνικών προϋπολογισμών να χρηματοδοτήσουν την αηφορία, την ε, προστασία του κλίματος και διάφορα τέτοια. Εάν βασιστούμε κυρίως στους, ε, στους, Ευρωπα... στους εθνικούς προϋπολογισμούς, θα καταλήξουμε σε μεγαλύτερη απόκληση ακόμα μέσα στην Ένωση και μάλιστα και στην ίδια την ζώνη ευρώ. Βλέπουμε τώρα στην οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη απόκληση και μέσα στη ζώνη ευρώ. Αυτό θέλουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό να δώσουμε υψηλότερη έμφαση στις κοινοτικές πολιτικές και να μετακινήσουμε ίσως ορισμένους εθνικούς στόχους προς την κατεύθυνση ευρωπαϊκών πολιτικών, κοινοτικών πολιτικών. Γιατί αυτό θα είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση όπου χρήματα που δαπανώνται στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα οδηγήσουν σε πιο συνεκτική και συγκεντρωτική προσπάθεια υλοποίησης των στόχων. Και αυτή λοιπόν ίσως είναι μια κατευθυντική σκέψη για το μέλλον. So, jetzt haben wir Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων. Πριν προχωρήσω να δώσω τον λόγο στον εισηγητή, θα ρωτήσω αν η Κομισιόν θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση, ενδεχομένως, γιατί εν τω μεταξύ έχουν τεθεί και διάφορες ερωτήσεις Ίσως θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες εξ αυτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί τη βάση των όσων άκουσα, έχω να σας πω τα εξής από δική μας πλευρά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη από όσα ελέγχθησαν ότι τονίστηκε στον προϋπολογισμό δεν καλύπτεται η στατική 2020. Υπάρχει στόχος. Θα πρέπει να πλαισιωθεί στον επόμενο προϋπολογισμό. Και έτσι να υπάρχει ένας γερός σύνδεσμος μεταξύ του σήμερα και του αύριο. Είδατε το σχετικό πίνακα που εκπονήσαμε. Φαίνεται εκεί πως έχει κατάσταση. Στη φάση προπαρασκευής του προεγγολισμού για τη χρήση 2011 γιατί υπάρχουν και άλλες πολιτικές της Ένωσης. Υπάρχουν προτάσεις για την οικονομική πολιτική θα πρέπει όμως αυτές τις προτάσεις να μετασχηματιστούν σε πράξη. <coughs> για όλες τις πολιτικές, πολιτική ανάπτυξη, εσωτερικών, όλα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Είτε έχει συνδέονται άμεσα με την οικονομία ή όχι. Δεύτερη παρατήρηση. με τους ίδιους πόρους. Είναι κάτι το οποίο απασχόλησε πολλούς από τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο. Είναι σημαντικό. στο εγγραφό μας την επόμενη εβδομάδα θα σας καλύψουμε. Ο, ο Επίτροπος, ο επικεφαλής υπηρεσίας μας, πρόεδρε κάποιες δηλώσεις το καλοκαίρι. Δημιούργησαν πολύ θόρυβο, αλλά δεν αφορά την αύξηση των πόρων αυτού το οποίο ελέγχθη, αφορά την αρχική μας φιλοσοφία όσον αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών. Άσχετα με το επίπεδο των πόρων, το οποίο είναι άλλη δύσκολη συζήτηση. θέμα των νέων ιδίων πόρων είναι κάτι το οποίο αφορά την αρχική προσέγγιση σε πρώτερη φάση των συνθήκων. Προοδευτικά ολιστήσαμε προς εθνικές συνεισφορές ανάλογα με το ΑΕΠ και φτάσαμε τελικά στο 70% εισφοράς του ΑΕΠ. Μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν θα υπάρξει θέμα αύξησης, ούτε δημιουργίας νέων πόρων. Απλώς θέλουμε να υπάρχει κάτι που είναι πιο συνεπές με την απαρχή της ευρωπαϊκής διαδρομής. να είναι ο κοινωνικό προπολογισμό πιο ουδέτερος. Αυτό για να έρθουν τυχόν παρεξηγήσει. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Τα όσα είπατε για τους ιδίους πόρους, βέβαια αυτά αναμέναμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ τουλάχιστον δεν ε, είχα καμία άλλη ε, σχετική αντίληψη. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε, ίσως μας ευνηδιάσετε του χρόνου. Εσύ τώρα, Σαλβαδόρ, σε παρακαλώ, την σύνοψη. Ναι, Πρόεδρε. Έχω συναντήσει ήδη τρεις γενικούς διευθυντές ε, αρμόδιους για τον προϋπολογισμό κατά τη θητεία μου εδώ και όλοι ο καθένας με τα καλά του και τα κακά του ο καθένας βοηθούσε όσο μπορεί και κανένας ποτέ δεν έδωσε καμία άμεση απάντηση ακριβώς και ο συνάδελφος που είναι σήμερα μαζί μας είναι πολύ σπουδαίος γενικός διευθυντής και ακολουθεί επομένως αυτήν την παράδοση. Στις ε, παρεμβάσεις. Να ξεκινήσω από την τελευταία, γιατί τα θυμάμαι καλύτερα αυτά τα οποία είπε. Ο Σκάλφιν. Πώς καλύπτονται από τον προϋπολογισμό τα flagships. Ένα συνάδελφο τη Γραμματεία μου είπε ότι στι 6 Δεκάτου έγινε η παρουσίαση τη πρωτοβουλία για την καινοτομία για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβησε μια υπέροχη εισήγηση όσον αφορά τις προκλήσεις για την καινοτομία και στην εισήγηση και παρουσίαση εκείνη για την καινοτομία Innovation Union λεγόταν ανακατεύονται εκεί διάφορα στοιχεία διάφορα στοιχεία ε, τα οποία αφορούν και τους τρεις στόχους την ευφύ ανάπτυξη, την βιώσιμη ανάπτυξη και έγινε μια εισήγηση αρκετά θολή σε σχέση με το από ποιο τμήμα του προεκλογισμού θα καλυφθεί αυτή η φλάξη. Υπάρχουν σημαντικέ μελέτε όσον αφορά την απασχόληση. Λέει για το 3% του ΑΕΠ, το οποίο αφιερώνεται στην ανάπτυξη. 3 εκατομμύρια 700.000 νέες ε, θέσεις εργασίας και το 2025 λέει για αύξηση 700 εκατομμυρίων το ΕΠ. Και διαβάζω, διαβάζω, διαβάζω και ψάχνω πού αναφέρει το πρωτοπολογισμός. Πουθενά. ή ε, κάπου θα υπάρχει. Δεν μπορεί όλη αυτή η υπέροχη έκθεση δεν περιέχει ούτε μία λέξη για τον προπολογισμό που θα καλύψει την Innovation Union. Νομίζω οποιοδήποτε από τους συναδέλφους βουλευτές θα συμφωνούσε ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αποφέρει έσοδα. Και άλλωστε η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με τις φλάξεις αλλά δεν μας λέει τίποτα για τον προπολογισμό. Για κοιτάξτε την πέμπτη σελίδα του κειμένου μου. Εκεί υπάρχει ένας πίνακας. Και εκεί αναφέρεται το 43% των δαπανών που θα καλύψει τις flagships. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε νέες δημοσιομικές προοπτικές για το 2020, αλλά θα πρέπει να αγνοήσουμε πάρα πολύ σημαντικού τομεί που οφείλει να καλύψει ο προπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν τώρα να κάτσουμε να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό ε, σε σχέση με τις νέες δημοσιογικές προοπτικές. Επομένως, η στρατηγική 2020 μήπως έχει την τύχη της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι των συναδέλφων και παρόντων και απόντων συμφωνούν. Θα πρέπει η στρατηγική αυτή του 2020 να προσαρμοστεί στις δημοσιομικές προοπτικές. Για θα πρέπει να παραδεχτούμε θα είναι, θα είναι αυτή η προσπάθεια όπως ήταν και η συνθήκη της Λισαβόνας. και αλλιώς θα πρέπει να δούμε πώς να το να κανείς για να εφαρμόσει την συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτές οι προοπτικές θα είναι η βάση για τη στρατηγική του 2020. Στη στρατηγική αυτή έχουμε και πολλές δαπάνες, ε, ζητήθηκε πιο σκληρή, πιο άγρια γραμμή, πιο καινοτόμα. Ο σημερινός προϋπολογισμός, όπως έχει, ταιριάζει στη νέα στρατηγική. Εμείς αυτό ζητούμε. Όμως πολιτικές μεταβλητές, πολιτική συγκυρία θα, θα δείξει κατά πόσον θα γίνει αυτό που θέλουμε, αλλά και το πώς θα δημορφωθεί ο προϋπολογισμός. Συγχρηματοδότηση μας είπε η κυρία Γένσεν. Βεβαίως, όλα αυτά είναι συγχρηματοδότηση. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι από σήμερα και στο εξή, ό,τι εντάσσουμε στη στρατηγική 2020 θα πρέπει να πληρεί το κριτήριο της συγχρηματοδότησης, που και αυτό θα γίνει αντικείμενο πάρα πολύ συναρπαστικής πολιτικής αναμέτρησης. Αυτό όπως θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Η συγχρηματοδότηση θα είναι η βάση πάσης πολιτικής. Ε, τι να κάνουμε, χρειάζονται κάποιε πολιτικέ αποφάσει που προποθέτουν κάποιο ρίσκο. Έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ σα τα είπα κύριε Πρόεδρε, τώρα θα πρέπει να τα πούν και οι, συνάδελφοι. Ήδη έχουν εκθέσει πάρα πολύ σημαντικέ ε, ιδέε και προτάσει. Και βέβαια θα πρέπει να ακούσουμε και τους ε, συναδέλφους που δεν ήταν σήμερα εδώ. Να πούν τη γνώμη τους και αυτοί σε μια άλλη μας συνάντηση. Να μας πούν τι πρεσβεύουν για αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με την παρέμβασή της μας διαφώτισε για το πώς βλέπουν την υπόθεση των ιδίων πόρων. Θα αντλήσουμε τα συμπεράσματά μας. Πάντως εγώ ακόμη αγνώ τι ορίζεται flagship και τι θα γίνει με την υπόλοιπη χρηματοδότηση που δεν προβλέπεται προς το παρόν. Σας είπα το Innovation Union ένα κλασικό παράδειγμα. Ό,τι πρωτοβουλία και να ψάξουμε, στο ίδιο θα καταλήξουμε. Και αυτό ακριβώς θα είναι η πρόκληση που η Επιτροπή μας, η Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, θα αντιμετωπίσει στους επόμενους μήνες. Το, χάσμα που υπάρχει μεταξύ προπολογισμού και στόχων. Ευχαριστώ καθώς και για τις προτάσεις και την πρόταση ιδιαίτερα να γίνει μια σύντομη σύνοψη και πάλι την... πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Βέβαια θα πρέπει να έχει σύντομο χαρακτήρα για να μην αρχίσουμε πάλι να συζητούμε και να θέλουν να λάβουν το λόγο και όλες και όλοι οι συνάδελφοι που δεν ήταν σήμερα παρούσες. Τώρα έχουμε έρθει στο υπαριθμόν 6 Υπάρχει κάτι που σας ενδιαφέρει υπό τα διάφορα. αν όχι, τότε ε, μόνο να πω το εξής, ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 28 Οκτωβρίου, Εθνική Ορτή, πέμπτη πρωί και πάλι. Αρχικά είχαμε βάλει και την πέμπτη απόγευμα, διότι είπαμε ότι ίσως θα πρέπει να γίνει εκείνη την ημέρα η ακρόασή μας. Τώρα την ακρόαση αποφασίσαμε να την κάνουμε τον Νοέμβρη, ώστε θεωρώ ότι η παρουσία σήμερα μου δείχνει ότι επουδενή δεν θα πρέπει να οργανώσω συνεδρίαση πέμπτη απόγευμα, διότι όχι μόνο δύο πολιτικές ομάδες λείπουν, υπάρχει και μια πολιτική ομάδα που έχει 13 τακτικά και 13 αναπληρωματικά μέλη, και που στην καλύτερη περίπτωση είχε παρόντα τέσσερα μέλη και τρεις αναπληρωματικούς. Και το πολύ πολύ να πω ότι ήταν και ο αντιπρόεδρος που ανήκει πάλι στην πολιτική μου ομάδα. Δεν ευθύνεται λοιπόν η σχετική απουσία εδώ μόνο στο ότι ορισμένοι βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό. Όποιοι θεωρούν ότι θίγονται αστιγούν από αυτά που είπα. Δεν ε, φίδομαι ούτε της ομάδας μου. Σαν ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Όπως είπα, την επόμενη φορά μια σύντομη σύνοψη, χωρίς να αρχίσει ξανά η μεγάλη ευρεία σύντηση. Ε, λοιπόν, 28 Οκτωβρίου το πρωί από τις 9 μέχρι την 12η και 30 μεσημβρινή και για το απόγευμα όχι. Καλή σας όρεξη.